Καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, με χαρά σας καλωσορίζω όλους εδώ στο πάνελ για τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και τη διαφορά μπορούν να προσφέρουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους στο πάνελ μας και τους καλωσορίζω, καθώς ιδιαίτερα ε, θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω την παρουσία των τριών ροβημένων με τον Σαχάροφ συναδέλφων και τον κύριο Λίμπο Ρούτσε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οποίο ευχαριστώ για την ευγενή συμμετοχή του στο πάνελ, καθώς και για τις ε, τελικέ του διατυπώσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να μιλήσω στα ελληνικά πλέον, δεδομένου ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, προάγουμε την ε, πολυγλωσία, την ε, διαφορά και έτσι προτιμώ να μιλήσω ελληνικά. Είμαστε όλοι μάρτυρες και θειασότες της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας. Είδαμε ότι τα μέσα επικοινωνίας με τη σύγχρονη τους μορφή δίνουν τη δυνατότητα σε προσωπικό επίπεδο μιας ελευθερίας στην έκφραση και επικοινωνίας των συμπολιτών μας, αλλά βλέπουμε ότι και σε επίπεδο συλλογικό δίνουν τη δυνατότητα σε κινήματα, σε οργανώσεις να επικοινωνούν και να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Είδαμε πόσο αυτό έγινε πράξη στον, στην Αραβική Άνοιξη, στο Arab Spring, όλοι εντυπωσιαστήκαμε από την απήχηση που είχε η οργάνωση μεταξύ των αγωνιστών, μεταξύ των διαφωνούντων ε, μέσω των μέσων επικοινωνίας. Σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση για αυτό το νέο θέμα, το οποίο έχει μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνική μας συμπεριφορά και στην πολιτική οργάνωση. Έχουμε στο πάνελ μας ε, ε, εξαιρετικούς ομιλητές. Καταρχάς, ο κύριος David John Collins,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 ο οποίος είναι blogger ε, ε, και ακτιβιστή για τα κοινωνικά δικαιώματα και προέρχεται από την Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Σε Σάκε, μέλος του Κοινοβουλίου, αγαπητή συνάδελφος. And, ε, Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και τις τοποθετήσεις τριών βραβευμένων με το βραβείο Ζαχάροφ ε, καταρχάς, ε, το, το ε, ε, είναι, την κυρία Ζάνα Λιτβίνα, Λιτβίνα, η οποία είναι δημοσιογράφος από την Λευκορωσία, την κυρία Χάουβα Ιμπραχήμ, που είναι από την Ιγυρία, νομικός, και θα έχουμε επίσης και τον κύριο Χέι Τζίγκεσμπέγκ, ε, ε, ακτιβιστή από την, ε, από την Κίνα. Θα δώσω το λόγο, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κόλινς. κύριε Κόλινς, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά περισσότερο, όπως και οι επόμενοι ομιλητές, για να μπορέσουμε να δώσουμε στο τέλος το λόγο και στο κοινό για κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις και ερωτήσεις. Ξεκινούμε από τον κύριο Κόλινς. Mr. Collins, the floor is yours. Thank you very much, and, and thanks for having me. Uh, real pleasure to be here, but το μικρόφωνο του μιλητή δεν είναι αναμένο. Καλημέρα σας. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ. Οι πραγματικοί όμως ήρωες της, ε, του αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης με τον κόσμο, αυτοί που κάνουν τη σκληρή δουλειά, είναι αυτοί που αναφέρατε ονομαστικά οι βραβευτέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Εμείς με εταιρείε όπως η Google έχουμε τεράστιους πόρους για τους ε, αγώνες αυτούς και μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά όταν κάποιος σε μια χώρα με κατασταλτικό, με αυταρχικό καθεστώς κινδυνεύει με την φυλάκιση, με τη στέρηση της ελευθερίας του, αυτός είναι ο πραγματικός αγωνιστής και πρέπει να τον τιμήσουμε. Ένα πράγμα δεν θέλω να πω, πολύ απλό, ότι για μας είναι επιχείρημα ε, και η έκφραση της ε, έκφραση μιας ηθικής διάστασης, η δυνατότητα της έκφρασης μέσω του ίντερνετ. Είναι τοποθέτηση δεοντολογική το να έχει κάνει τη δυνατότητα της πρόσβασης και της επιλογής στην έκφραση που θεωρεί ο ίδιο ότι τον εκφράζει καλύτερα. Ανεξάρτητο του τι θέλει να πει μια κυβέρνηση ή ένα κρατικό μηχανισμό να του επιβάλλει, να του βάλει στο στόμα και επιπλέον ε, την εποχή αυτή της ελεύθερης online έκφρασης και της ε, ε, τεχνοκρατικής διαμόρφωση ελευθερίας τη έκφρασης Καλό είναι να μην λησμονούμε αυτή τη διάσταση. Γι' αυτό η Google με τόσο μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό. Εμείς εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό για τη λειτουργία μας από την ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Δεν θα μπορούσα να ισχυριστώ κάτι αντίθετο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για μας θέμα δεοντολογίας να μπορεί κανείς να εκφραστεί ελεύθερα. Ένα παιδί στο Μπαγκλαντές, το οποίο πριν από 10-15 χρόνια δεν θα είχε καν πρόσβαση σε μια εγκυκλοπαίδεια. Γιατί μπορεί να μην έχει κοντά του, να μην έχει εύκολη πρόσβαση βιβλιοθήκη, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε ένα εργαστήριο και να δουλεύει συνέχεια. Ε, το ίντερνετ του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, δυνατότητες ανήκουσε στο παρελθόν. Δυστυχώς όμως πολλές είναι οι αρχές, πολλές είναι οι κρατικές εξουσίες ανά τον κόσμο που παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία. Και δυστυχώς πριν από 8-9 χρόνια ακόμα είχαμε σχετικά λίγες εταιρείες ε, κυβερνήσεις στον κόσμο που επέβαλαν φίλτρα στο ίντερνετ και έλεγχαν την πρόσβαση. Τώρα όμως είναι πολύ περισσότερες. Εδώ και 5-6 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών των κυβερνήσεων και των κρατικών μηχανισμών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε δυστυχώς ε, ότι ναι μεν αναπτύσσεται αυτός ο αγώνας μέσα του ίντερνετ, κερδίζει. Πολλοί από τους εδώ παρόντες ε, μιλάνε πολύ ανοιχτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου ο αγώνας αυτός δεν στέφεται με επιτυχία είναι αποτυχημένος και αν κοιτάξουμε γύρω-γύρω μπορούμε βεβαίως να επιλύψουμε ευθύνες, αλλά επίσης πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πέραν της δυνατότητας της έκφρασης ανά τον κόσμο και στις δυτικές δημοκρατίες που θεωρούμε ότι είναι λιγότερο κατασταλτικές από τις υπόλοιπες περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση. Βέβαια το ενδιαφέρον για το Google και τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ε, από τους κρατικούς μηχανισμούς ενισχύεται, όπως ενισχύεται η παρεμπόδιση και το φιλτράρισμα ε, των πληροφοριών που διαθέτουν τα ε, site αυτά ή στους σελίδες αυτές. Σας διαβεβαιώ βέβαια ότι το Google θα συνεχίσει τον αγώνα, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει και θα σας υπενθυμίσω γιατί το πράττουμε. Σας, το, σας υπογραμμίζω λοιπόν το πράττουμε και υπενθυμίζω το πράττουμε για λόγους ακριβώς αυτής της διοντολογίας που ανέφερα νωρίτερα και γιατί θέλουμε ο κάθε ένας να μπορεί να διεκδικεί το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορία που τον ενδιαφέρει, σε ελεύθερη έκφραση και πάντα μέσα στα όρια του δικαίου. Και εμεί θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό εκείνων που αποδίονται σε αυτόν τον αγώνα. Thank you very much for this uh, presentation and contribution. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Κύριο veteran of several ε, human rights λοιπόν πολλών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Um. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είναι σημαντικό με το διαδίκτυο είναι ότι ε, από την αρχή ξεκίνησε σαν ένα αποκεντρωμένο, ε, ολοκληρωμένο ε, σύστημα και βοήθησε την επικοινωνία και νομίζω ότι ε, και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας δίνει τη δυνατότητα ε, ομότιμης επικοινωνίας, μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, καθώς επίσης να οργανώνουμε και να κινητοποιούμε ε, ανθρώπους. Πολύ πιο εύκολα αυτό γίνεται επιγραμματικά παρά offline. Επίσης βοηθάει την ροή των πληροφοριών και επομένως παρακάμπτεται με τον τρόπο αυτό ε, η προσπάθεια αρχών εξουσιών να ε, ξεπεράσουν ε, και να περιγράψουν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται μια ελεύθερη ανταλλαγή περιεχομένου. Τώρα υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα σε αυτό που είπα μέχρι τώρα και τις ε, εθνικές ραδιοτηλεοπτικές αρχές. Το περιεχόμενο είναι διαφορετικό, οι αρχές είναι διαφορετικές και κατά κανόνα ε, χρησιμοποιούνται για εθνικούς λόγους. Ε, βεβαίως ε, στο διαδίκτυο ε, ξεκίνησαν τα πράγματα διαφορετικά ε, και ξέρετε για να κάνουμε μια σύγκριση ένας μηχανικός αυτοκινήτου φτιάχνει το αυτοκίνητο όσο και αν το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να τρέξει περισσότερο ή ανεξάρτητα με το σε ποια κατεύθυνση τελικά θα πάει το ε, διαδίκτυο, όπως έχει ήδη υποθεί, ε, δεν είναι ουδέτερο. Εξαρτάται από το ποιος το χρησιμοποιεί, τι τεχνολογία χρησιμοποιεί, ποια υποδομή και πώς λειτουργεί αυτή η υποδομή και επομένως ε, από εκεί εξαρτάται εάν θα είναι δύναμης καλού ή δύναμης κακού το διαδίκτυο. Ε, απ' την άλλη πλευρά μπορούμε, όπως είπα και προηγουμένως, να κινητοποιήσουμε κόσμο, να δούμε τι κάνουν ε, κατασταλτικές κυβερνήσεις, ε, τι κινήσεις ε, κάνουν ε, και βεβαίως συνδυασμένο το διαδίκτυο με την κινητή τηλεφωνία και τις δυνατότητες αποτύπωσης εικόνας που δίνει η κινητή τηλεφωνία, πραγματικά οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν χρειάζεται επίσης ε, οργάνωση, δηλαδή είδαμε και στις τελευταίες κινητοποιήσεις ότι αυτοί οι οποίοι κινήθηκαν και οργανώθηκαν μέσω του διαδικτύου δεν ήταν μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων ή ακτιβιστές ε, κτλ. Και στη Μέση Ανατολή Μάλιστα, διαπίστωσα ότι το παραδοσιακό κίνημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν συμμετέσχει καταρχήν ε, στις κινητοποιήσεις αυτές. Ε, φαίνεται ότι ε, ήταν λίγο δύσκολο να ξεκινήσει και να ταυτοποιηθεί με αυτό το κίνημα το οποίο ξεκίνησε online. Όσον αφορά τώρα τον ουδέτερο χαρακτήρα του διαδικτύου, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα στην οποία ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι περιεχόμενο θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Και γενικώ οι κυβερνήσεις ε, δεν ε, αρέσκονται σε αυτό και βεβαίως ε, οι κατασταλτικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες καθόλου δεν θέλουν κάτι τέτοιο και προσπαθούν μέσω τεχνικών εμποδίων, μέσω νομοθετικών προσκομμάτων να σταματήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, η, την άλλη πλευρά βεβαίως είναι γεγονός ότι στην Κίνα ας πούμε έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό ίντερνετ το οποίο ε, δημιουργεί προστατευτικό τείχος απέναντι στην χρήση του ίντερνετ και επομένως δεν έχουν πρόσβαση στο ε, κανονικό ε, τείχος. Από την άλλη πλευρά βεβαίως μπορεί να βρεις οτιδήποτε ε, στο διαδίκτυο, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές και από εγκληματίες και από ακραίες ιδεολογικές οργανώσεις, από ναζί, από οτιδήποτε, από ανθρώπους που προσπαθούν μέσω εγκληματικών ενεργειών να αποσπάσουν χρήματα The French government called for it at G8 in Paris early this year. Και βεβαίω σε πολλέ ε, περιπτώσει ε, ε, γίνεται μια προσπάθεια χειραγώγηση τη πληροφορία που διαχέεται μέσω του διαδικτύου και στη Ρωσία. Έχει γίνει αυτό και στην Κίνα και, και σε άλλε χώρε. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να λειτουργήσει το ίντερνετ όχι σαν ένα φόρουμ ελεύθερων ανταλλαγών αλλά σαν ένα μέσο χειραγώγηση και ε, προσπαθούν ε, βεβαίως ε, να μετα το ίντερνετ σε ένα είδος δορυφορικής τηλεόρασης. Ε, δηλαδή στη Συρία, ακόμα και αν έχεις καλωδιακή τηλεόραση, τα ίδια θα βλέπεις, ενώ και σε άλλες χώρες μπορεί κανείς μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης να πιάσει όμως τα κανάλια τα οποία ελέγχονται στην ουσία. Ε, και επομένως με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να δυναμητιστεί το ελεύθερο δημοκρατικό ίντερνετ το οποίο έχουμε εμείς εδώ. Ε, υπάρχουν βεβαίως ε, και κάποια προβλήματα επικοινωνίας ε, και προβλήματα γνώσης της πληροφορίας και διάδοσης της πληροφορίας που τώρα πλέον τον 21ο αιώνα έχουν γίνει κομμάτια των, της, του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αλή Νοβρούζοφ, τώρα έχετε τον λόγο. Κύριε Νοβρούζοφ από το Αζερβαϊτζάν. Θα ξεκινήσω Λέγοντα το εξή. Με ονομάζετε blogger, αλλά προέρχομαι από μια χώρα που το ίντερνετ δεν είναι ιδιαίτερα προχωρημένο. Είμαστε 9 εκατομμύρια Αζέρι και μόνο το 1 τρίτο του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Και από όλου αυτού του χρήστες, μόνο το 20% έχει πρόσβαση σε υψηλή ταχύτητα σε ευρυζωνικό ίντερνετ. Οι υπόλοιποι είτε δεν το χρησιμοποιούν, είτε το χρησιμοποιούν ε, σε μια ε, πρωτόγονη μορφή. Ακόμα λοιπόν και στον Πακού που είναι το, η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν αυτή και όπου έχουν γίνει πολλές ε, προσπάθειες να αναπτυχθούν οι υποδομές. Οι υποδομές που έχουμε είναι πεπαλαιωμένες και οι ταχύτητε του ίντερνετ είναι 2-3 ΜΜ το λεπτό, κάτι το οποίο είναι γελίο για τα δικά σας δεδομένα και είναι και πάρα πολύ ακριβό για να το συγκρίνουμε τόσα στοιχεία εδώ. Άρα λοιπόν στο Αζερβαϊτζάν, ο μέσος χρήστης είναι κάτοικος πόλεως, με σταθερό εισόδημα και βέβαια άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του. Στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή βρίσκεται η αιχμή της μάχης που δίδεται στο Αζερβαϊτζάν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και να σας εξηγήσω τι συνέβη. Και πώς συνέβη αυτό σε μια χώρα όπου οι υποδομές μας, επαναλαμβάνω, είναι πολύ παπαλαιωμένες. Πώς έγινε το ίντερνετ το βασικό εργαλείο. Πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο τρέχον πολιτικό σύστημα της χώρας, το οποίο είναι απολυταρχικό, παρόλο που είμαστε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως επίσης και του ε, ε συστήματος ε, γειτονία ε, ε, με τις ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θέση των του βαθμολογικού πίνακα των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα έχουμε καταλάβει τη θέση 152. Και πριν από δύο χρόνια ήμασταν στο 113. Αλλά καταλαβαίνετε πως όχι μόνο δεν πάμε καλά, αλλά είχαμε και ραγδαία πτώση αυτά τα τελευταία χρόνια. Το Αζερβαϊτζάν πρέπει να πω ότι έχει τις χειρότερες φυλακές για δημοσιογράφους στον κόσμο και δεν υπάρχει εκδότης μεγάλης εφημερίδας που να μην έχει πέρασει από τη φυλακή. Μάλιστα είχαμε και μία εποχή που δύο εκδότες ήταν ταυτόχρονα φυλακισμένοι. Η κυβερνήση έχει ε, κλείσει τους αντικαθεστατικούς τη δυνατότητα να μιλήσουν στις πλατείες, στα πανεπιστήμια, στους ραδιοσταθμούς. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν αποτύχει. Άρα λοιπόν οι, ναι, οι ομάδες των νέων που είναι και πιο φιλελεύθεροι έχουν ε, στραφεί στο ίντερνετ για να προωθήσουν ε, και τον αγώνα που κάνουν και την προσπάθεια για να χαίρουν των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ έντονη αντίφαση μεταξύ του τι συμβαίνει στην καθημερινότητα της ζωής του Αζερβαϊτζάν, όπου τα πάντα βρίσκονται υπό έλεγχο, που ακολουθείται μια πολύ συγκεκριμένα ρουτίνα με απόλυτο έλεγχο της καθημερινής ζωής, αφενός και από την άλλη έχουμε ε, τη ζωή στο ίντερνετ, η οποία είναι ελεύθερη, ανοιχτή, τεχνικά τουλάχιστον, και όπου έχουμε οδηγηθεί μέσω όλων αυτών ε, ε, ε, συσσωρευμένων πιέσεων να προκηρύξουμε την δημοκρατία του ίντερνετ, του facebook. Δηλαδή ζούμε στη δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν με σοβιετικό ρυθμό ζωής και στη δημοκρατία του Facebook όπου είμαστε ελεύθεροι, μιλάμε και αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Αν εξετάσουμε το πώς έτυχε να είναι ελεύθερο το ίντερνετ σε μια χώρα όπως το Αζερβαϊτζάν, γιατί μας έχει απασχολήσει. Η μεν κυβέρνηση είναι καταπιεστική, αλλά φαίνεται να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτα αλήθεια, γιατί ε, σε τεχνικό επίπεδο δεν έχουμε ούτε λογοκρισία, ούτε φίλτρα, ούτε τύχη, αλλά η κυβέρνηση καταπιέζει πάρα πολύ όσους είναι ακτιβιστές στο ίντερνετ, γιατί κατανόησε η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες ή τις ε, δράσεις που κάνουμε στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να στρέφεται προς μεθόδους ε, παλαιού τύπου, που είναι η τις δρασεις που κανουμε στο ιντερνετ με αποτελεσμα να στρεφεται προς μεθοδους παλαιου τυπου που ειναι η φυλακιση ε, ο ξυλοδαρμή. Το 2009 Δύο ακτιβιστές από το ίντερνετ φυλακίστηκαν γιατί ανέβασαν ένα σατυρικό βίντεο. Και αν μπείτε στο Google θα το δείτε. Τους λένε donkey bloggers. Και έκανε ό,τι μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έκανε ό,τι μπορούσε και ο κύριος Μπούζεκ, νομίζω και εσείς βοηθήσατε και προσπαθήσατε να απελευθερώσετε αυτούς τους δύο bloggers, τους donkey bloggers. Αυτοί απελευθερώθηκαν και μπήκαν άλλοι δύο θέσεις στη φυλακή. Η Διεθνής Αμνηστία έχει ε, μία, ένα κατάλογο με πέντε χώρες όπου ό,τι σχολιάσει στο ίντερνετ μπορεί να σε στείλει στη φυλακή. Κίνα, Βιετνάμ, Συρία και Αζερβαϊτζάν είναι τα μέλη του καταλόγου αυτού. Δύο λοιπόν είναι ο κύριος Μπαρσαβαλάν και ο Μπασταρ Χατζήρ που έχουν μπει ε, φυλακή. Ο δεύτερος ε, σπούδασε στο Χάρβαρτ και γύρισε στη χώρα του να κάνει κάτι για την πατρίδα του. Και φυλακίστηκε για τη δράση του. Ως συμπέρασμα θέλω να πω το εξής. Το ίντερνετ για την κυβέρνησή μας μοιάζει με, με το αμερικανικό τραγούδι που λέει γύρισε η γάτα. Ο κύριος Τζόνσον προσπαθούσε να διώξει τη γάτα και η γάτα όλο γύριζε στο σπίτι. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση. Και το είπε και ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης. Το ίντερνετ είναι μια μαύρη γάτα, άτιμη που μπορεί να υπερπηδήσει οποιοδήποτε φράχτη και να μπει στου καθενό στο σπίτι χωρί να τη ανοίξει την πόρτα. Για την κυβέρνησή μα λοιπόν είναι αυτή η μαύρη γάτα το ίντερνετ. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να τη διώξουν. Mm. Όμως δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα ως συμπέρασμα να πω πως αυτή τη στιγμή οι αντιφρονούντες, οι κυβερνού αντιφρονούντες του Αζερβαϊτζάν συνεχίζουν τον αγώνα. Και χτες είδα την έκθεση όπου η δημόσια τηλεόραση η δημόσια τηλεόραση του Αζερβαϊτζάν συκοφάντιζε αυτό τον blogger που πήγε στην Ευρώπη και προσπαθεί να αμαυρώσει τη φήμη της χώρας του. Συκοφαντική. Συκοφαντική εκστρατεία λοιπόν εναντίον blogger, ε, χώρο που όπω σα είπα ανήκει και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, αλλά αποτελεί και τμήμα των χωρών στην εταιρική σχέση γειτονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, και τώρα η σύνθεση κυρία Σάκε. Ενεργό μέλο Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Μάσκη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την, τον Πρόεδρο, την Πρόεδρο και όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρία, σε αυτή την οργάνωση που πάνω απ' όλα εξασφάλισαν την παρουσία τόσων πολλών από τόσα πολλά έτη βρεβευθέντων με, ε, με το Ζαχάροφ ε, αγωνιστών. Αισθάνεται κανείς μικρός μπροστά στα δικά σας ονόματα, μπροστά στη δική σας παρουσία. Και πίσω από εσά βεβαίω, πίσω από τα ονόματά σα υπάρχουν τόσοι άλλοι άγνωστοι που δεν ξέρει κανεί το όνομά του, αλλά που και αυτοί έχουν αγωνιστεί πίσω σα. Και πιστεύω ότι έτσι διευρύνονται και οι κύκλοι, ε, οι ομόκεντροι κύκλοι του αντικτύπου που μπορεί να φέρει η δουλειά σα. Στα μέσα μαζική ενημέρωση λοιπόν ε, ιδιαίτερα, αλλά και στην, ε, στα θέματα τη νεολαία, τη παιδεία, όπου δραστηριοποιούμε, υπάρχουν πολλά να πούμε όπως και για το εθνές εμπόριο που εντάσσεται στο θέμα αυτό. Τεχνολογία λοιπόν, ανθρώπινα δικαιώματα. Ζούμε σε εποχές τεραστίων αλλαγών, τρομερών αλλαγών. Εάν ε, θυμηθούμε την περίοδο των εκλογών στο Ιράν πριν από δύο χρόνια, το 2009, όπου ήταν τόσες χιλιάδες εκείνοι που κατέβηκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν την ψήφο τους, να αναγνωριστεί η ψήφος τους. Τώρα το, το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει ένα λεγόμενο ίντερνετ χαλάλ, ε, καθαρό δηλαδή, σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις αρχές με λογοκρισία δηλαδή. Το ίδιο η Κίνα, το ίδιο οι άλλες χώρες ε, και όπως και χώρες της Βόρειας Αφρικής που είδαμε πόσο μεγάλη σημασία μπορούσε να δραματίσει στο διαδίκτυο στις χώρες αυτές, αλλά και στις δικές μας κοινωνίες ε, παρά ίσως ε, τις ε, χωρικές αποστάσεις που τους χωρίζουν, οι άνθρωποι μπόρεσαν, οι πολίτες μπόρεσαν να ενωθούν, μπορούν να αμφισβητήσουν την εξουσία και να φέρουν σημαντικές αλλαγές στις δημοκρατικές κοινωνίες και τις δικές μας δημοκρατικές κοινωνίες αλλά και σε εκείνες που γνωρίζουν περισσότερη καταστολή. Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σαφώς έχει προχωρήσει και έχει προχωρήσει online εγώ το κόμμα από το οποίο προέρχομαι ονομάζεται D66 που είχε την, ε, είχε την πρόθεση όταν ξεκίνησε με το πρόγραμμά του πριν από δύο χρόνια να διεκδικήσει ως ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση στο ίντερνετ. Κάποιοι βέβαια αντέδρασαν λέγοντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει υποβάθμιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων εν γέννη, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα υπό την έννοια της πρόσβασης στην ε, πληροφορία αλλά και τη κατάρριψης των ταμπού σε κοινωνίε όπου είναι πιθανόν αδύνατο ή ε, πολύ δύσκολο να συστήσει κανείς φερειπίν τη σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών. Ε, μπορεί να τεθούν ζητήματα έξω από τον έλεγχο των αρχών. Πρόσβαση λοιπόν στις νέες αρχές, στις νέες τεχνολογίες, δικαίωμα του συνέρχεστε, καθώς στις κοινωνίες μας η στη σύγχρονη κοινωνία η καταγραφή ε, και η τεκμηρίωση δεδομένου ότι υπάρχουν παντού κάμερες ε, χειρός και μη ε, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ευχερής πλέον. Βέβαια αυτό ίσως είναι και δυσμενής εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν, πριν έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εργαζόμουν στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για την ε, Ιουγκοσλαβία, για την και παρακολουθούσα τις μελέτες, τις ε, δηλώσεις των μαρτύρων, μελετούσα δηλαδή τα κείμενα που ερχόντουσαν ε, και τις καταθέσεις των μαρτύρων και ήταν, θυμάμαι, πολύ δύσκολο να βρούμε φωτογραφικό υλικό για να τεκμηριώσουμε κάποια δήλωση κάποιο ισχυρισμό. 15-20 χρόνια πριν μόλις και είχαμε τόσο λίγο εποπτικό υλικό στη θέση μας, είχαμε μόνο, γραπ... δηλώσεις. Τώρα έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε να κερδίζουμε από την εμπειρία ένας του άλλου. Πολλοί άνθρωποι έχουν ε, υποστεί βασανισμούς για να αποκαλύψουν το ε, κωδικό που χρησιμοποιούν για πρόσβαση σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης ε, όπως το Facebook και Το ίδιο στην Τινησία ξέρουμε ότι η δικτατορία του Μπεναλή προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την υψηλή τεχνολογία για να έχει πρόσβαση στους προσωπικούς λογαριασμούς ε, email και τα λοιπά των αντιφρονούντων. Το ίδιο και με τη Συρία για να επανέλθω σε αυτά που έλεγε ο συνάδελφος, ε, από το, ο συναγωνιστής από το Αζερβαϊτζάν, υπήρξαν προσπάθειες για παρακολούθηση μέσω του διαδικτύου της κινήσεως και των κινήσεων των ε, αντιφρονούνταν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ε, προσπάθειες και από τα Ηνωμένα Έθνη για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων τόσο στο, στη Συρία όσο και στο Ιράν και την Μπαχρέιν, όπου ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από τους πολιτικούς κρατουμένους στο Ιράν, παραδείγματι, αντιμετωπίζουν ε, σαν εις βάρος τους πιστήριο τα ίδια του τα email, δηλαδή έχει πρόσβαση η αστυνομία στα email και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του. Το ίδιο όμω βλέπουμε να συμβαίνει και στον Ηνωμένο Βασίλειο ει βάρο κάποιων υποπτών τρομοκρατών. Έτσι λοιπόν, για να καταλήξω από ό,τι, πρέπει, από φαίνεται πρέπει να τελειώνω, πρέπει να μην υπερβάλλουμε ω προ την επιβολή νομοθετικών ρυθμίσεων. Πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, οι πολίτε, την δυνατότητα μόνοι του να δρουν και να κάνουν τι επιλογέ του. Μπορεί να υπάρχουν διάφορε πλατφόρμε, αλλά υπάρχουν κάποια θεμελιώδη στοιχεία τη δημοκρατία Υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση για τη δημοκρατική εποπτεία, την εποπτεία ότι τηρούνται δημοκρατικά όνες δημοκρατίας δηλαδή, αλλά και η διάκριση των εξουσιών και η δυνατότητα τη πρόσβαση στο ίντερνετ, χρειάζεται η διαφάνεια, χρειάζεται διαφάνεια για πλευρά των επιχειρήσεων για να ξέρουμε ποιο εξάγει τι σε ποια κοινωνία, ώστε να μην ε, συμβάλλουμε άθελά μας στην ε, ενίσχυση καθεστώτων αυταρχικών εις βάρος των πολιτών τους. Αυτά πολύ ξεκάθαρα νομίζω σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε τις κινήσεις του εμπορίου, του διεθνούς εμπορίου και ταυτόχρονα ε, θα πρέπει όταν μελετούμε τις νέες τεχνολογίες να αναλογιζόμαστε τι είδους θετικές αλλά και αρνητικές κυρίως επιπτώσεις μπορεί να έχει αξιοποίησή τους στόχοι στρατηγική, στόχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρήση των ε, τεχνολογιών ε, από εταιρείε πολλέ φορέ εδρεύουσε στη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέματα τα οποία μα απασχολούν. Θα ήθελα επίση να πω ότι το, ίντερνετ έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και έχει αλλάξει πολλά στη ζωή μα, αλλά δεν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα Έχουμε και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες με τους θυμημένους, με το βραβείο Ζαχάροφ, την κυρία Λετβίνα του 2004. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Για πέντε λεπτά. Ε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω ρώσικα. Τα πρώτα μου λόγια είναι λόγια ευχαριστίας για τη δυνατότητα που μου δώσατε να λάβω το λόγο σε αυτό το χώρο που για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί αντιμετωπίζετε τα προβλήματα όχι μόνο του επαγγελματικού μου κλάδου αλλά και της χώρας μου και στα πλαίσια αυτών των προβλημάτων, δηλαδή της ανάπτυξης του ίντερνετ και της καταπίεσης αυτού, πρέπει να τονίσω το εξή στις μη δημοκρατικές χώρες είναι η μοναδική δυνατότητα που έχει ο κόσμος να λάβει πληροφορίες, να αναμεταδώσει πληροφορίες γιατί στα μη δημοκρατικά καθεστώτα αυτό που κάνουν ότι κρατάνε την εξουσία στα χέρια τους, μονοπολούν την πληροφορία και πιέζουν μέσω της δικής τους προπαγάνδας και για τον απλό κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσανατολιστεί. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στην ίδια του τη χώρα ο λαός. Δεν μιλώ για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Με το συγκεκριμένο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στη Λευκορωσία βλέπουμε ως πολύ θετικό φαινόμενο το γεγονός πως υπάρχει μια ιδιαίτερη ζήτηση ε, πληροφορίας η οποία δεν έχει λογοκριθεί, η οποία είναι ελεύθερη. Και ίσως αυτό είναι το στοιχείο το οποίο ε, δίνει τη δύναμη στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και τους υποστηρίζει γιατί κατανοούν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους και τη σημασία που έχει όχι μόνο το να βρουν αλλά και να διαδώσουν τις πληροφορίες. Αυτό το κάνουν μέσω του ίντερνετ στη χώρα μας και η σημασία του είναι η ακριβώς δυνατότητα αναμετάδοσης ειλικρινούς πληροφορίας. Βεβαίως η κυβέρνηση είναι κατά ε, της ε, ε, κατά της διεύρυνσης πρόσβασης στο ίντερνετ. Ε, εμείς αντιδράσαμε σε κάποιες προσπάθειες που γίνανε από την κυβέρνηση να χειραγωγήσουν το ίντερνετ και αυτή τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες που ε, προσφέρονται στη χώρα μας θα πρέπει να ε, έχουν μεταφραστεί και να έχουν καταχωρηθεί από την κυβέρνηση. Και για να πας και σε ίντερνετ καφέ πρέπει να δείξεις ταυτότητα. Διαφορετικά δεν μπορείς να μπεις και να ζητήσεις έναν υπολογιστή και να βγεις στο ίντερνετ. Δηλαδή, σου ζητάνε τουλάχιστον να δουν το διαβατήριό σου ή την εσωτερική σου ταυτότητα. Καταλαβαίνετε τι στιγμέ ζούμε και υπάρχουν και μαύροι κατάλογοι που υπάρχουν 30 ε, περίπου ε, Μίντια έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο. Ε, δεν μιλάω για ακραίες, ε, για ακραία μίντια. Θα έλεγα ότι είναι ε, προωθημένα. Είναι ο, ο Παρτιζάν για τα παράδειγμα και μία ακόμα σειρά πηγών ενημέρωσης που έχουν μπει σε μία μαύρη λίστα και η πρόσβαση στα site αυτά απαγορεύεται και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση ούτε από κυβερνητικά κτίρια, ούτε από κυβερνητικά ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια ε, ελέγχου ε, του ίντερνετ, παρόλο που εξακολουθεί το ίντερνετ να παραμένει ως μια ζώνη ελευθερίας. Αυτό λοιπόν ε, κάνει το ίντερνετ και μας βοηθάει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην διεθνή κοινότητα. Γιατί για παράδειγμα γίνονται κάποιες δίκες Ξέρετε τι γίνεται με τον κύριο Μπελιάτσκι. Μόνο online έχουμε κάποια δημοσιογραφικά κείμενα που μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τι γίνονται στη δίκη του. Το δεύτερο το οποίο καλύπτει το ίντερνετ και είναι πολύ σημαντικό ε, στην Λευκορωσία είναι η κινητοποίηση. Μετά από τις τελευταίες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ε, είδαμε τι σημαίνει πώς να κινητοποιείς τον απλό πολίτη. Ποια είναι η δυνατότητα που έχει ο λαός να μαζευτεί, να συγκεντρωθεί και να εκφραστεί μέσω της και ήταν πραγματικά λαμπρά τα αποτελέσματα. Και κάναμε κάποιε διαδηλώσει χωρίς αρχηγού, χωρί σημαίε, χωρίς λάβαρα. Ήρθε ο κόσμο. οι άνθρωποι οι οποίοι ε, με μία ψυχή και με μία πεποίθηση αποφάσισαν, συναντήθηκαν σε ένα σημείο και σιωπηλά, χωρίς αρχηγούς και κόμματα, κατέβηκαν στις πλατείες και άρχισαν απλώς να χειροκροτούν. Και ο απεχθής τρόπος με τον οποίο τους έδιωξαν, ο βίος και βάναυσος τρόπος με τον οποίο από φόβο βέβαια οι κυβερνητικές υπηρεσίες τους καταδιώκουν, γιατί βέβαια η κυβέρνηση φοβάται ε, την χειραφέτηση αυτή, αποδεικνύει ε, πόσο δυνατό είναι το ίντερνετ, γιατί στην Λευκορωσία η αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους, που είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γίνεται μέσω ίντερνετ. Δηλαδή μαζεύουμε υπογραφές, μαζεύουμε ε, χρήματα για οικογένειες των φυλακισμένων, ε, για όσους έχουν υποφέρει από κάποιο καταπιστικά μέτρα. Όλα αυτά μέσω ίντερνετ. Και πρόσφατα, αυτό το οποίο πιο πολύ μας ανησυχεί, μας τρομάζει, είναι το γεγονός πως η χώρα μας έχει πέσει σε μια τεράστια απομόνωση. Για παράδειγμα, εγώ που προσπαθώ να μπω σε κάποια κοινωνικά δίκτυα μέσω ίντερνετ, για να δώσω κάποιες ελπίδες και να κάνω κάποια, να, να δώσω μία ανάσα γιατί πραγματικά η νέα τεχνολογία δίνει αυτή την ελπίδα. Ε, φοβάμαι και φοβάμαι ότι η χώρα μου θα περιέλθει πάλι σε αυτή την προηγούμενη κατάσταση της κλειστής επικράτειας, ε, όπου οποιαδήποτε ε, δημοκρατική αλλαγή δεν θα γίνει γιατί μεταρρυθμίσεις χρειάζονται πληροφορίες, χρειάζεται πρόσβαση των πολιτών, των συμπολιτών μου στο ίντερνετ. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις δυσκολίες ε, ελεύθερης πληροφόρησης και χρήσης του ίντερνετ, ερχόμαστε σε μια άλλη πύρο στην Αφρική, η, η βραβευμένη με το γραφείο Ζαχάροφ το 2005, η κυρία Ιμπραχήμ, από την Ιγυρία, δικηγόρος και δραστήρια στα, στην πρόσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, θα πάρει το λόγο. Κυρία Ιμπραχήμ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και η αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίως δε η. Ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με προσκάλεσε εδώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Κάνετε εξαιρετική ε, δουλειά και πραγματικά ε, στηριζόμαστε και σε εσά. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Και μετά βεβαίως θα απαντήσω και στις ε, ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές γλώσσες υπάρχει η γλώσσα της τεχνολογίας και υπάρχει και η γλώσσα της επιστήμης. Νομίζω ότι οι γυναίκες θα πρέπει, κυρίως δε γυναίκες από τον αναπτυσσόμενο χώρο, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε αυτό το νέο κόσμο και ευχαριστούμε που μας βοηθάτε όσον αφορά την ε, τεχνολογία γενικότερα και την, την τεχνολογία της επικοινωνίας ειδικότερα. Δεύτερον, θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο σχετίζεται με την ε, επιρροή των γυναικών σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέλλον για το οποίο θα είμαστε περήφανες, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναμειχθούμε με όλα τα στοιχεία και τις εκφάνσεις αυτής της νέας τεχνολογίας. Θα ξεκινήσουμε από χαμηλά θα ξεκινήσουμε από τα χωριά μας, γιατί ξέρετε εμείς στις δικές μας περιοχές, στα δικά μας χωριά, για πολλά χρόνια έχουμε αγωνιστεί για να σταματήσει ο αναλφαβητισμός και για να έχουν και γυναίκες πρόσβαση στην, ε, στην ε, εκπαίδευση. Εμείς θέλουμε να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή, να δώσουμε δύναμη σε αυτούς που δεν έχουν δύναμη, να ε, βοηθήσουμε. Γιατί, ξέρετε, Ακόμα και το τηλέφωνο είναι δείγμα ε, εξουσίας. Ε, η γυναίκα πρέπει από το δικό της το χωριό να μπορεί ε, να τηλεφωνήσει, θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να δημιουργήσει δυνατότητες για ε, να προοδεύσει για να κάνει εμπόριο. Ε, δηλαδή ε, μια γυναίκα που θα είναι ας πούμε μια γυναίκα η οποία θα πουλάει οτιδήποτε στην αγορά θα μπορεί με το τηλέφωνο να μάθει την τιμή αυτού του προϊόντος. Θα πάρει τηλέφωνο την αγρότησα που βρίσκεται στην αγρικία της και θα τη ρωτήσει τι τιμή χρειάζεται για το προϊόν αυτό. Ξέρετε, σε ένα, παλιό, σε ένα μικρό χωριό, σε ορεινή περιοχή, ε, είδα μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία απαντούσε στο τηλέφωνο και πραγματικά ε, μου είπ, αισθάνθηκα ε, αισθάνθηκα πολύ περίεργη και της είπα πώς τηλεφωνείς, ε, βάζεις ε, τους αριθμούς ε, και είπε ναι αλλά επειδή εγώ δεν έχει αριθμούς στο τηλέφωνο μου, έχει γράμματα και επειδή δεν τα ξέρω έχω, έχω βάλει τα παιδιά μου και μου λένε ποια νούμερα θα πρέπει να χτυπήσω. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ακόμα και για αυτή την απλή δουλειά πρέπει κανείς ε, να είναι εκπαιδευμένος. Επομένως η εκπαίδευση, η έξοδος από την άγνοια είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την απλή τεχνολογία για να προχωρήσουμε. Ε, και βεβαίως ο δρόμος για το μέλλον περνάει μέσα από το δρόμο της αξιοπρέπειας που δεν σχετίζεται ούτε με το φύλλο μας, ούτε με το ε, χρώμα του δέρματός μας. Πρέπει για το μέλλον να καταλαβαίνουμε πλέον την γλώσσα της τεχνολογίας, τη γλώσσα της επιστήμης που είναι κοινές γλώσσες. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιμπραήμ κύριος Σιγχέγγε από την Κίνα. Ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, μετά την ε, Αραβική Άνοιξη αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το ίντερνετ για να κινητοποιήσει τους πολίτες, πόσο σημαντικό όπλο για μια επανάσταση μπορεί να είναι. Ε, δεν είναι πολύ καιρό τώρα που αντελήφθησαν τη σημασία του ίντερνετ οι Κινέζοι πολίτες και έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο ίντερνετ. Συχνά μάλιστα μπορούν να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις τους να δώσουν να κάνουν παραχωρήσεις. Και με τον ε, Τσάι που είχαμε πρόσφατα στην επικαιρότητα, μπόρεσε η πίεση της κοινή γνώμης να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του. Τώρα όμως προσπαθούν οι αρχές πάλι να βρουν κάποιο λόγο για να τον συλλάβουν. Υπάρχει όμως μεγάλη δικτύωση. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι συνέβαλαν, δορίζοντας μάλιστα εκατομμύρια, ε, εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν για να βοηθήσουν στον αγώνα αυτό. Είναι λοιπόν το ίντερνετ μεγάλο εργαλείο, σπουδαίο εργαλείο για να μπορεί ο λαός να εκφράσει τη φωνή του. Οι δυτικέ εκείνες εταιρείε που ίδρυσαν το ίντερνετ βεβαίως έχουν συμβάλει με τον τρόπο αυτόν ιδιαίτερα, έχουν βοηθήσει τους λαούς, αλλά δεν είναι τα πάντα θετικά πρέπει να πούμε διότι παραδείγματι Η Κίνα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που επέβαλε ε, τη λογοκρισία της στο ίντερνετ. Οι χώρες, δυτικές χώρες ε, με το Google, με το Yahoo, έχουν χάρη σε αυτές τις ε, πληροφορίες που συλλέγονται, προσφέρει στην κυβέρνηση της Κίνας στοιχεία για τη δραστηριοποίηση των πολιτών της. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν μας βοηθάει καθόλου. Δεν βοηθάει καθόλου αυτού του θαραλέου που θέλουν να σηκώσουν, να υψώσουν τη φωνή τους για να εκφράσουν ελεύθερα τι ε, απόψει τους. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα ως προς τις χώρες και τις εταιρείε από, το δυτικό κόσμο που δεν έχουν ισοδηληφθεί σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει κατάχρηση των πληροφοριών που εξασφαλίζονται μέσω του διαδικτύου, μέσω της νέας τεχνολογίας από κυβερνήσεις ε, αυταρχικές. Ο κόσμος δεν έχει πραγματική ελευθερία πάντα, ε, δεν προσφέρει το ίντερνετ πραγματική ελευθερία. Ε, πολλές φορές οι κινέζικες αρχές με τη στήριξη, με την αρρωγή δυτικών επιχειρήσεων μπορεί να επιβάλλει βαριά καταστολή και με παρακάλεσαν οι συναγωνιστές μου να το υπογραμμίσω αυτό ιδιαιτέρως. Γιατί υπάρχουν δικτατορίες οι οποίες με τη βοήθεια αυτών των επιχειρήσεων έχουν παρεμποδίσει την ελεύθερη έκφραση των αγωνιστών. Ελπίζω λοιπόν οι χώρες αυτές της Δύσης, οι κυβερνήσεις αυτές του δυτικού κόσμου να προχωρήσουν προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω όπως βλέπουμε τώρα. Φερρυπίν, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Με πολύ προσοχή χειρίζονται το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Κίνα ε, με το γάντι θα έλεγα, παραβλέποντας τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η δε κινέζικη κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να εισακούσει εκκλήσεις από τις δυτικές χώρες. Οι Κινέζοι αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, κλιπαρούν να ακουστεί η φωνή τους, αλλά κανείς δεν τίνει ευήκον ους. Και η κυβέρνηση της Κίνας τους σφαλίζει το στόμα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι αφόρητη. Αυτό που μου έχουν ζητήσει συναγωνιστέ μου να σας πω από την Κίνα είναι ότι η κινέζικη κυβέρνηση δεν πρόκειται ούτως ή άλλως να διασώσει τι ευρωπαϊκέ χώρε όσο και αν αυτέ το ελπίζουν διότι τι θεωρεί εχθρό απλώ και μόνο. Δεύτερον, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδει αξίε του ανθρώπου ελπίζω να μην λησμονηθούν από τι χώρε του δυτικού κόσμου. Ελπίζω να μην χάσουν αυτό το ιδεώδε, δηλαδή στο βωμό τη ευημερία των business, των επιχειρήσεων με την Κίνα. Γιατί ξέρω βεβαίω ότι θέλετε να έχετε τι εμπορικέ συναλλαγέ, αλλά μην λησμονείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και με παρακάλεσαν οι σύντροφοι από την Κίνα να τα πω αυτά. Βεβαίω δεν μπορώ εδώ να εκφράσω, να ισχυριστώ ότι εκφράζω ή ότι εκπροσωπώ ολόκληρο τον κινέζικο λαό, αλλά μπορώ να σα πω ότι είναι πολύ γενναίο ο κινέζικο λαό, ότι είναι πολύ γενναίοι όλοι αυτοί οι αγωνιστέ ε, που ε, εδώ και ε, χρόνια έχουν αγωνιστεί και συνεχίζουν να αγωνίζονται και να ελπίζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αγωνίστηκαν και οι αγωνιστές της Αραβικής Άνοιξης. Παρακαλώ λοιπόν να μην κοιτάτε μόνο τους, μακροπρο... τους βραχυπρόθεσμους στόχους, αλλά να κοιτάτε και προς το μέλλον. Μην ξεχνάτε, Φερρυπίνο, ότι στην Αραβική Άνοιξη έγιναν ε, σφάλματα γιατί δεν είχαν γίνει αντιληπτοί οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πολιτών των κρατών αυτών της Βόρειας Αφρικής. Οι δυτικές χώρες δεν είχαν αντιληφθεί ποια ήταν η κατάσταση επακριβώς και παρέβλεψαν πολλά προβλήματα. Καλό λοιπόν είναι να κοιτάξετε να καταλάβετε τι συμβαίνει και στην Κίνα, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν διδραματίσετε ρόλο εσείς δραματικό, ε, ουσιαστικό, θα χάσετε την αγάπη, θα χάσετε το θαυμασμό που τρέφει για σας ο λαός της Κίνας. Γιατί ο λαός της Κίνας προσβλέπει με θαυμασμό στο δυτικό κόσμο, στο δυτικό πολιτισμό και στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες αυτού του κόσμου. Όμως θα τους χάσετε εάν δεν τους στηρίξετε και πρέπει να βοηθήσετε έτσι ώστε να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ να κάνουν μια πρώτη αντίδραση σύντομη, ενός λεπτού, ε, στα αυτά που ήδη τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπαν οι laureates. Ε, στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας. Αυτή τη στιγμή θα ρωτήσω τα μέλη του πάνελ αν θέλουν να αντιδράσουν. Ο κύριος Κόλλινγκς ήδη θέλει να κάνει μια πρώτη παρέμβαση. Κύριε Κόλλινγκς. One minute, please. Thank you very much. I, I think like all of, all of the people in... Νομίζω πως όπως και όλοι οι υπόλοιποι ευχαριστάμενοι εντυπωσιάστηκαν από τα όσα άκουσαν και εμψυχώνονται και εμπνέονται και πρέπει να σα πω ότι στην Κίνα ποτέ δεν παραδώσαμε πληροφορίες περί, περι, ε, περι για τους χρήστες στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλες εταιρείε, αλλά εμείς πήραμε την απόφαση αυτή πριν ξεκινήσουμε την προσφέρουμε τις υπηρεσίες πριν από κάποια χρόνια και είπαμε πως δεν θα το κάνουμε. Και πέρσι ε, δεν κάναμε πλέον και λογοκρισία στην ε, αναζήτηση ε, στο, στο engine search στην Κίνα με τις γνωστές επιπτώσεις. Νομίζω πως οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν τη μάχη εναντίον του ίντερνετ. Άρα λοιπόν θα πρέπει όσοι βρισκόμαστε εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι υπόλοιποι, να συνεχίσουν τον αγώνα υπέρ ανθρώπων που είναι πολύ πιο άτυχοι από ότι εμείς. Άλλος κανείς? No. Okay, okay. Eh? At the end of... No. No, okay. I thought maybe the previous speakers were, were also going to be first. Um, no, just very briefly. I... Στα γρήγορα να σας πω πως είναι πολύ χρήσιμο και βεβαίως επιβεβαιώνει και την μάχη που δίνω σε αυτό το κοινοβούλιο είναι η αξιοπιστία της Ευρώπης που διακυβεύεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ξέρετε πως οι ιδέες μας εξάγονται ε, και ξαφνικά πολλές φορές οι άλλες κυβερνήσεις, ε, οι κυβερνητικές εταιρείες, οι κρατικοί οργανισμοί, η αστυνομία και όσοι συνεργάζονται με αυτά τα κατα καθεστώτα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να περιορίσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία. Και Ξέρετε πως κυκλοφορεί αυτή η ιδέα πως υπάρχει και η νόμιμη παρακολούθηση. Πότε δηλαδή μπορεί η αστυνομία να παρακολουθεί τις ιδιωτικές συνομιλίες ε, των ανθρώπων. Όταν για παράδειγμα εξαφανίζεται ένα παιδί ή αγνοείται η χιονού ενό σκιερ ε, σε μια χιονοστιβάδα. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το διαφορετικό πλαίσιο σε περιπτώσεις που ισχύει το κράτος δικαίου, όπου η αστυνομία σε μια ε, δημοκρατική ελεύθερη χώρα με διάκριση εξουσιών ε, χρησιμοποιεί το σήμα του κινητού για παράδειγμα για να εντοπίσει κάποιον και το τι σημαίνει αυτό σε κράτη όπου δεν ισχύει το κράτος δικαίου, όπου χρησιμοποιούν το σήμα του κινητού για να βρουν σε ποια γωνία, σε ποια πλατεία ποιας πλατείας έχουν μαζευτεί 10 άτομα για να φωνάξουν για τη δημοκρατία. Άκουσα και τα όσα είπε η κυρία Ιμπραήμ για το πόσο σημαντικό είναι να έχει πρόσβαση στο ανοιχτό ίντερνετ και πόσο θα πρέπει να δίνεται αυτή η δυνατότητα σε όλους και κυρίως στις γυναίκες. Νομίζω αυτό το σχόλιο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη δεόντως. Το λόγο θα δώσω το λόγο στον καθηγητή ε, κύριο Πουσιβίλη από το Διεθνές Κέντρο για τις σειράξεις και τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές ε, τις ε, τόσο ε, σημαντικές παρεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητούμε την χρήση της τεχνολογίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου δεν χρειαζόμαστε πλέον, δεν, δεν χρειάζεται πλέον να περιοριστούμε ε, όταν μιλάμε για κινήματα ανεξαρτησίας. Ε, δεν χρειάζεται πλέον να προστρέχουμε στην ε, Γαλλική Επανάσταση. Νομίζω πλέον ότι μπορούμε να μιλάμε για την επανάσταση της τεχνολογίας και την πρόσβαση στην τεχνολογία που είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του κάθενό μηδενό εξαιρουμένου σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας. Πολλοί μεταξύ ημών ε, έχουν ε, ε, ζήσει την σιωπηρή συνεργασία με τους παρόχους ε, των ε, δικτύων γνωρίζουμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές, γνω, πολλές χώρες έχουν αλλάξει την νομοθεσία τους έτσι ώστε ε, η εξουσία να μπορέσει να παρέμβει σε την διάδοση της πληροφορίας ε, φτάνουμε ε, σε έναν ε, κόσμο που το σημείο αυτό πρέπει να προσεχθεί γιατί μπορεί να αποτελέσει σημείο χειραγώγησης και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει άμεσα να αντιδράσουν. Πρότασή μου λοιπόν είναι να σκεφτούμε το ενδεχόμενο της ελεύθερης ροής πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο και να το βάλουμε, λέω, στην ε, διακήρυξη των, ε, διεθνή διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε ε, να σηκώνουμε κόκκινη κάρτα σε όποια κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Και τώρα από την Ουγκάντα έχουμε την πρέσβυρα Μίρια Μπλακ. Please, your proposals. Γεια σας πρόταση παρακαλώ. We have 50 minutes for interaction. Sorry, I have not asked for the floor, Madam Chair. Κυρία Πρόεδρε, δεν ζήτησα το λόγο εγώ. Δεν ζήτησα το λόγο. Oh, okay. Please. Can you introduce yourself, please? Yes, yes. Θα μας πείτε το όνομά σας. Είναι Ήρθον Σίκμαν από τη Σερβία. Εκπροσωπώ την, ε, το κίνημα αντίστασης ε, κατά τον Μιλόσεβιτς. Και τώρα εκπροσωπώ τον τομέα κατάρτισης της οργάνωσης. Καταρτίζουμε ανθρώπους από πολλές χώρες, από τις Μαλδίβες, την Γεωργία, της, ε, πρόσφατα, από τη Γεωργία πρόσφατα και από την Αίγυπτο και από το Λίβανο. Εμείς δεν ασχολούμαστε με πολιτικά θέματα. και πιστεύω ότι υπάρχει μια παγίδα σε αυτά τα νέα μέσα. Δηλαδή, ε, είναι ένας ε, εικονικός κόσμος και στον εικονικό κόσμο μπορείς να κερδίσεις τον αντίπαλό σου, αλλά τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο, όπως εξήγησαν και οι πανελίστες μας. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να μείνει, δηλαδή ένα εργαλείο και σαν εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Θα προσπαθήσω όμως να ε, ρίξω λίγο διαφορετικό φως. Ε, ας πούμε ότι είναι σε πρωτόλια κατάσταση το διαδίκτυο στην ε, I Το διαδίκτυο στη Σερβία ε, και ε, επομένως ε, είναι σημαντικό βεβαίως που μπορούμε να, βλέπουμε πράγματα στο διαδίκτυο, αλλά εάν κανείς κάθεται στην καρέκλα του και παίζει στο διαδίκτυο και δεν κατεβαίνει στις πλατείες για να διώξει το Μιλόσεβιτς, τότε εκεί αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. 40.000 ε, άνθρωποι ε, ξεκίνησαν μια ολόκληρη επανάσταση και στη Λιβύη έγινε αυτό και αλλού. Νομίζω γενικά ότι θα πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν την μη βίαιη δράση ε, έτσι ώστε να μην έχουμε ματοχυσίες όπως ας πούμε στη Λιβύη ή στο Αφγανιστάν παλιότερα και ελπίζουμε να μην το δούμε και στη, να συμβαίνει στη Συρβία. Αυτά. Στη Συρία. Ευχαριστώ. Very much. Thank you. Please. Could you introduce yourself, please? Yeah. My, name is Sipin Hua, λέγομαι. και εδώ και 20 χρόνια περίπου ασχολούμαι με, την, ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ και 27 χρόνια ασχολούμαι με το ίντερνετ. Ενδεχομένως ε, είμαι από τους πιο ηλικιωμένους ε, όσον αφορά το, το διαδίκτυο. Έχω υπάρξει και computer manager για κάποιο διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ σημαντικό εργαλείο το διαδίκτυο. Θα ήθελα να εκφράσω μια ανησυχία και από τον πολιτικό κόσμο και από τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να στηρίξει ε, το δημοκρατικό κίνημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην ε, Κίνα. Ξέρουμε ότι πριν από μερικά χρόνια η Γιαχού ε, ήρθε σε επαφή με την ε, κυβέρνηση της ε, Κίνας και με τον τρόπο αυτό φυλακίστηκαν κάποιοι αντιφρονούντες και εδώ ο κύριος Γιανχού επίσης φυλακίστηκε με τον ίδιο τρόπο κάποια στιγμή πολλά χρόνια πριν ε, η Google ανοίξει, πριν σπάσουν οι λογαριασμοί της Google από ε, κάποιους, ε, μερικοί ακτιβιστές μας μας είχαν πει ότι είχαν υποστεί πειρατεία οι λογαριασμοί τους. Και Ε, υπάρχουν εταιρείες όπως η Cisco ας πούμε στην ε, Δύση που βοηθούν ε, την κινέζικη κυβέρνηση εξάγοντας τεχνολογίες και δυνατότητες πειρατείες και όταν έχει όλα τα στοιχεία η αστυνομία μπορεί μέσω της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε μισή ώρα να έχει πιάσει τον αντιφρονούντα. Ε, και αυτού του είδους η τεχνολογία βεβαίως έχει εισαχθεί από την Δύση. Γι' αυτό λοιπόν η δυτική βιομηχανία, οι δυτικέ κυβερνήσεις, οι δυτικοί, ε, ε, ε επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί αυτή η τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούς τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του κακού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Μπαζίλια. Πολύ σύντομα. Ο πόλεμος, γιατί για πόλεμο πρόκειται, διεξάγεται σε δύο μέτωπα. Στο μέτωπο του γραπτού και στο μέτωπο της τεχνολογίας. Για το γραπτό λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία, άτυπη γιατί έτσι δουλεύουμε, που έχουν, στην οποία έχουν αποδειθεί οι πρόσωποι της κοινωνίας ε, των βραβείων Ζαχάροφ με μια έκκληση την οποία έχουν μέχρι τώρα υπογράψει πέντε από τους βραβευθέντες και που θα απευθύνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλοι. Ζητούμε λοιπόν να μην υπογράψει το Κοινοβούλιο το άκτα, το κείμενο αυτό που είναι θεμελιώδη σημασία για το ίντερνετ του αύριον. Ένα κείμενο βεβαίως με σημασία εμπορική, αλλά με τεράστιες επιπτώσεις και αντίκτυπο στην ελευθερία του ή στην ελευθεροτυπία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντισταθεί όχι μόνο στη διατηφίση των επιδιωκομένων μέσω του ΑΚΤΑ, αλλά και στο κείμενο το ίδιο. Ξέρουμε επιβεβαίως ότι οι βουλευτές εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό, ωστόσο και καθώς εγώ παρακολουθώ την ομοπαραγωγική διαδικασία μέσα από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μετατρέπονται σε νόμο οι προθέσεις, όμως δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε διακήρυξη προθέσεων ή σε, απλές, ε, σε απλά ευχολόγια ή χάρτες δικαιωμάτων. Ίσως η λύση θα ήταν να πούμε, και αυτό βέβαια δεν θα πιστέψω το λέει κάποιο που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλη τη ζωή, ε, αλλά θα ήταν το πιο σωστό να πούμε ότι βγάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από το κείμενο και αφήνουμε μόνο τη διάσταση τη αγορά. Τότε δεν θα έχει κανένα νόημα βεβαίω. Ενώ τώρα έχουμε αυτού οι οποίοι διεκδικούν ένα ίντερνετ ανοιχτό, συμμετοχικό, με streaming, με ε, μοίρασμα με συμμετοχή δηλαδή των πάντων και από την άλλη τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός ίντερνετ που απαρτίζεται από διαφορετικά ίντρανετ που θα μας επιβάλλουν οι χώρες. Δηλαδή αύριο θα έχουμε μπροστά μας ένα ίντρανετ ευρωπαϊκό που δεν θα έχει καμία επικοινωνία με το αμερικανικό ίντρανετ το οποίο θα είναι θωρακισμένο ε, και κλειστό προς τα έξω. Γι' αυτό θέλουμε να σταματήσει η λογοκρισία στο open source. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί μας δίνουν χρήματα για να βρίσκουμε μέσα αντί να αντιμετωπίσουμε την καταστολή. Από την άλλη όμως μας κλείνουν την πόρτα της τεχνολογίας και του open source. Είναι παράλογο αυτό και πιστεύω ότι ένα κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει κάτι το πολύ σημαντικό, κάτι το πολύ ουσιαστικό στο τομέα αυτό. Υπογραμμίζω λοιπόν την έκκληση προς το Κοινοβούλιο. Μην υπογράψετε το ΑΚΤΑ. Μία συμφωνία που έχει τύχει τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεως δεν έχει θέση σε ένα αντιπροσωπευτικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Προσθέσατε μια νέα διάσταση στη συζήτησή μας. Και ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο, κύριε, παρακαλώ. Ε, je suis, ε, un militant Είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, αλλά είμαι και στο Βέλγιο, ε, μια και είμαι πρόσφυγας από τη χώρα αυτή. Ε, σήμερα το πρωί δεν είχαμε εκπρόσωπο του Ιράν που να έχει κληθεί. Σήμερα το απόγευμα όμως είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έχουμε και την κυρία Σάκη, η οποία είναι μέλος της Σχετικής Επιτροπής και γνωρίζει τα θέματα του Ιράν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά εξηγήσατε το τι γίνεται ε, και ποια είναι η λυπηρή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Για τον φίλο από την ε, Google έχω δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία. Θα συμφωνήσω. Καμιά φορά όμω κρύβει και κινδύνους. Για παράδειγμα, δεν προσέχει ιδιαίτερα στον περσικό κόλπο. Ε, δεν αναφέρεται στον περσικό κόλπο ως περσικό, αλλά ως αραβικό κόλπο. κόλπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική σύραξη αυτή η λέξη, οπότε ίσως η Google θα πρέπει να προσέξει πώς τον ονομάζει. Δεν έχει αλλάξει το όνομα στα Ηνωμένα Έθνη και γιατί αλλάζετε εσείς το όνομα του περσικού κόλπου που και τον κάνετε αραβικό κόλπο, δεν κατάλαβα ποτέ. Δεύτερον, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρώπη αποφάσισαν να επιβάλλουν κυρώσει στην Ιρανική κυβέρνηση. Ρωτώ την Google, μπορείτε κι εσείς να κόψετε στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Ε, για παράδειγμα, για το ποιο έχει παράγει πληροφορίες και τις έχει βάλει στο ίντερνετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ε, που έγιναν, θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Όχι. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Κόλλιντς και μετά στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ, αν επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Κύριε Κόλλινς. Um, um, Ευχαριστώ πολύ για το εκ του Google. Δεν έχω μιλήσει πολλές φορές σε δημόσια πάνελ, αλλά ξέρω πάντα ότι ο κόσμος έχει πολλές ερωτήσεις και σωστό είναι αυτό. Για τον εκπρόσωπο του, για τον κύριο που μίλησε από το Ιράν, δεν θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ δύσκολο να προσφέρουμε υπηρεσίες σε μια χώρα όπου τις, διεθνείς, τις διευθύνσεις ε, ICP της ελέγχει η κυβέρνηση. Άρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε ε, υπηρεσίες από ε, ίσο προς ίσο δεδομένου αυτού του ελέγχου. Ο τρόπος με τον οποίο ονομάζονται οι διάφορες περιοχές, ε, οι γεωγραφικές ονομασίες δηλαδή, φαντάζομαι ότι υπονοείται ότι πρόκειται για το Google Maps ως υπηρεσία. Πολύ ευχαριστώ να το ξανακοιτάξω. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, περιοχές του κόσμου που εκφράζονται διαφωνίες προς το όνομα που δίνεται. Πολύ ευχαριστώ να το κοιτάξω λοιπόν και να έρθω σε επαφή μαζί ε, στη συνέχεια. Και επίσης θέλω να πω ότι η σύγκρουση με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν νομίζω περιγράφηκε από μένα νωρίτερα ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Οι τελευταίοι πιστεύω θα ήμασταν ε, που θα ήθελαν να ζητήσουν συνεργασία οι αρχές του Ιράν ούτως ή άλλως. Αλλά εν πάση περιπτώσει το συζητάμε και διμερώς αν θέλετε. Μια ιδιαίτερη έκκληση πάντως ε, για μέτρα και πρωτοβουλίε θα μπορούσε να ανάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συμφωνήσω μαζί σα για τι εξαγωγέ τεχνολογία που αναφέρθηκε νωρίτερα. Θα μπορούσα λοιπόν να προτείνω και ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπήρξε μια ε, πρόταση πλευρά τη ε, Ολλανδία για την απαγόρευση τη ε, τεχνολογία ελέγχου. Επίσης η πρόταση για την περίληψη της πρόσβασης στο διαδίκτυο τον, ε, στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, αλλά ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε σαν πρώτο βήμα να αντιμετωπιστεί και μέσα από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, διότι το, η λογοκρεσία χρησιμοποιείται ως εμπορικός φραγμός από ορισμένε χώρες, από ορισμένε κυβερνήσεις και θα μπορούσαμε και μέσω αυτού να το, ε, να, το καταπολεμήσουμε. Ο κύριος Πόλιουφα τα έχει το λόγο. Πούρεφατ. Ένα-δύο σημεία μόνο. Ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο άρθρο 19 του του συστήματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουμε το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Και άρα πιστεύω ότι υπάρχει εγγύηση από τις υφιστάμενες, από τα υφιστάμενα νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις το δικαίωμα της πρόσβασης στο ίντερνετ. Το να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών συζήτηση για πρόταση για υιοθέτηση μέτρων και δικαιωμάτων πρόσβασης στο ίντερνετ θα ήταν αποτυχία καταδικασμένο εξ αρχής και πάντως το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήγουμε θα ήταν μάλλον ελάχιστα ικανοποιητικό δεν έχουμε πλέον το ρεύμα που είχαμε όταν μπορούσαμε να περάσουμε τόσες προτάσεις όπως δεκαετία του 90. Τώρα μάλλον είναι αρνητική η συγκυρία και ιδιαίτερα χώρες οι οποίες υπεστήριζαν τα ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Αφρική επί παραδείγματι, τώρα τα καταψηφίζουν και θα ε, ήταν μάλλον άφρον κίνηση να προταθεί κάτι τέτοιο μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη. Πάντω ήταν καλό να το διερευνήσουμε, γιατί Cisco Φερρυπίν ξέρετε ότι η τεχνολογία ε, των επικοινωνιών έχει εξαχθεί ε, έχουμε, σε σχέση με την Κίνα όλα αυτά αλλά και με την Nokia και με τη Siemens είχαμε προτάσεις για εξαγωγές σε χώρες όπως το Ιράν και έτσι θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουν αλλάξει σε ένα βαθμό στάση αυτές οι επιχειρήσεις. Απέριψαν δηλαδή μια σειρά από ε, συμβάσεις που τους είχαν προταθεί όπως άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα σεμινάριο τις οποίες όμως ανέλαβαν στη συνέχεια επιχειρήσεις από την ίδια την Κίνα και έτσι ε, ίσως μετακινείται το βάρος και το σημείο εστίασης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οι τεχνολογίες που αξιοποιούν χώρες ε, αυταρχή, με αυταρχικά καθεστώτα, βλέπουμε ότι τώρα αξιοποιείται ε, όχι ως ένα τυχαίο υποπροϊόν, αλλά ως κύριο προϊόν, ως προϊόν ανάπτυξης, ως αντικείμενο ανάπτυξης από επιχειρήσεις σοβαρές, έστω και μικρές, στην Ιταλία, τη Γερμανία και Ελλαχού και που προσπαθούν να πουλήσουν ως κύριο προϊόν, ως κύρια υπηρεσία αυτήν την τεχνολογία. Μικρέ επιχειρήσει υπογραμμίζω, όχι τεράστιε πολυεθνικέ που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κανεί. Μικρέ επιχειρήσει που θα μπορούσε πολύ εύκολα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στοχεύσει και να περιορίσει τη δράση του. Είναι γνωστό και αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά το προϊόν που παράγουν, πού πηγαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρικέ σχέσει με την ε, Bloomberg ε, και, τη, και που, συλλέγουν, καταγράφουν αυτές τις πληροφορίες. Είναι εύκολο λοιπόν να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν τη σχετική τεχνολογία. Αυτά τα οποία ακούσατε νωρίτερα δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση με τα όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ. Ναι, θα, είμαι... θα είμαι πολύ σύντομη. Χαίρομαι που εκπρόσωπος της ε, Google στηρίζει το ελεύθερο ίντερνετ και άλλες ε, πρωτοβουλίες ε, γιατί εμείς θεωρούμε σαν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Θέλουμε λοιπόν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά να έχουν συνείδηση αυτών των πραγμάτων. αλλά ε, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν εταιρείε και όπως η Cisco η οποία ε, κάνει τέτοιου είδους, ε, πουλάει τέτοιου είδους τεχνολογία. Πάντως πρέπει να σας πω ότι μήνες πριν την επίσημη δήλωσή σας εμείς ήδη από τους ακτιβιστές μας ε, ε, ξέραμε ότι η κινέζικη κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει hackers για να, ε, για, για να σε, να σπάσουν λογαριασμούς αντιφρονούντων. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που τώρα μιλάτε υψηλόφωνα για το θέμα αυτό και λέτε ότι όντως υπήρξε, υπήρξε πρόβλημα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς τα ξέραμε αυτά ένα χρόνο ολόκληρο. Ε, πριν ξεκινήσουν, ε, πριν μιλήσετε εσείς και η Yahoo επίσης ε, αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό η Yahoo συνεργάστηκε με την κινέζικη κυβέρνηση και έστειλε τελικά πολλούς αντιφρονούντες στη φυλακή και πήρε περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια σαν αποζημίωση. Και βέβαια το μόνο που ήθελαν στην ουσία όταν ξεκίνησε, όταν ακούστηκε το ζήτημα ήταν απλώς να προστατεύσουν τη φήμη τους και όχι να βοηθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι που με απασχολεί. Πρέπει να σας πω ότι όταν η μυστική αστυνομία στην Κίνα με συνέλαβε, οι κινέζικες αρχές μου είπαν θα μπορούσες να έχεις κερδίσει δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή εάν ε, μας βοηθούσες να χτίσουμε αυτό το firewall ε, στην ε, Κίνα. Και μου είπαν, ορίστε ακόμα και με μεγάλες εταιρείες μας βοηθούν. Επομένως και επομένως ε, γιατί δεν μας βοηθάς και εσύ. Εμάς, ε, ε, σας λέω για μία ακόμα φορά, μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Ευχαριστώ. Thank you so much. Uh, to for... Ευχαριστώ πολύ για τις καταπληκτικές σας παρεμβάσεις. Νομίζω ότι η δουλειά μας τώρα ξεκινάει και από τα ίσα είπατε όλοι, νομίζω πως είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρο τον κόσμο, τους νέους ηλικιωμένους. Έχουμε θέματα πολιτικά, εμπορικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξωτερικής πολιτικής. Όλα άπτονται αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να σας καλέσω όλους, από όπου και αν προέρχεστε, από ΜΚΑ, ομικρόν, από κυβερνητικές οργανώσεις και κυρίως όσοι έχουν βραβευτεί, να συνεργαστούν μαζί μας για να διατυπώσουμε κάποια στρατηγική ε, online ελευθερίας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σφαιρική, συνολική και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο και στον Αντιπρόεδρο, κύριο και για τα τελικά συμπεράσματα, τα τελικά σχόλια από τα όσα άκουσε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ρόδη. Συζητάμε εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης και την τεχνολογία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία σκέψης, έκφρασης, πληροφορίας, είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω πως από τα δικαιώματα αυτά απορρέουν τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι, για παράδειγμα, το δικαίωμα του συνέρχεσθε, ε, του συνδικαλίζεστε. Ε, είτε αυτό είναι κάποιο πολιτικό κόμμα, είτε συνδικάτο ή κάποια ένωση ε, επιχειρηματιών. Είναι λοιπόν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία όπως ακούστηκε εδώ στην αίθουσα, έχουν περιγραφεί πάρα πολύ σε πάρα πολλές δηλώσεις. Έχουμε βέβαια τις δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε τις ευρωπαϊκές ε, και σε άλλα μέρη του κόσμου. Όμως, και θα ήθελα εδώ να απηχήσω ότι είπε ο κύριος Μπάζελ σήμερα το πρωί, το ευρωπαϊκό μοντέλο μας είπε ότι έχει σπάσει. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όμως σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου έχουμε παραβιάσεις και παραβιάζεται συχνά και στην Ευρώπη. Μιλήσατε για την Ουγγαρία. Ναι, ο νόμος περί τύπου στην Ουγγαρία όντως πρόκειται για μια παράφορη ε, καταπάτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου. Το ίδιο συνέβη στην Ιταλία. Το σκάνδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή ε, έχει ε, ταράξει το Ηνωμένο Βασίλειο με την ε, εταιρεία του κυρίου Μέρντοκ. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου παραβιάσεις και εμείς πρέπει να τις ε, αποτρέπουμε. Η τεχνολογία εξελίσσεται, μεταλλάσσεται. Οι φίλοι στη Σερβία αναφέρθηκαν την εποχή που το ίντερνετ ήταν στα σπάργανα και τον ρόλο που έπαιξε την, ε, στο κίνημα της αντιπολίτευσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να σας πω τη δική μου ιστορία. Όταν ήμουν ακτιβιστής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξόριστος δεκαετία του 70 και του 80, δεν είχαμε ούτε ίντερνετ, ούτε κινητά. Ούτε φαξ δεν είχαμε τότε, οπότε τι κάναμε, τυπώναμε. Είτε στην Ολλανδία, είτε στη Βιέννη, είτε στο Μόναχο, τυπώναμε ε, σε, σε τυπογραφία και περνούσαμε τα έντυπα αυτά λαθρέα από Τσεχοσλοβακία και από άλλες χώρες. Μετά εμφανίστηκαν ε, τα φωτοτυπικά, τα φαξ. Τα πράγματα ε, άλλαξαν, διευκολύνθηκαν. Είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να οργανώσεις κινήματα όλων των ειδών με τη νέα τεχνολογία μέσω κινητών, με το ίντερνετ. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θα είχε γίνει ο σοβιετικός τύπου κομμουνισμός εάν είχαμε τότε, πριν από 25 χρόνια πριν, τέτοια τεχνολογία στην α, διάθεσή μας. Θα είχε επιβιώσει ο κομμουνισμός ή θα είχε η τεχνολογία οδηγήσει σε μια πιο γρήγορη κατάρρευση του συστήματος. Να, μια ερώτηση η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί. Η τεχνολογία λοιπόν τα, οι μοντέρνοι τρόποι επικοινωνίας έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στο να ανοίγουν κλειστές κοινωνίες σε αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Νοβρούζοφ, στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν, δεν έχουν όλη πρόσβαση σε υπολογιστές, στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει στο Αζερβαϊτζάν και νομίζω και από την Αφρική θα μας απαντήσουν ότι η κατάσταση είναι παρόμοια, δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Τι χρειάζεται λοιπόν έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να έχουν περισσότερη πρόσβαση. Γιατί είναι σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όπως είπε και η κυρία Ιμπραχήμ, είναι σημαντικό για την παιδεία και βέβαια για τις γυναίκες. Οι γυναίκες για να χειραφετηθούν πρέπει να απελευθερωθούν από κάποιους παραδοσιακούς τρόπους ζωής που επιβάλλει περιορισμούς όλων των ειδών. Ο κύριος Νοβρούζοφ είπε πως υπάρχουν δύο ειδών κοινωνίες η κοινωνία στην οποία υπάρχει πρόσβαση και η κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει πρόσβαση και όπου ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τα επίσημα ΜΜΕ, μια και δεν έχει τα τεχνικά μέσα ε, για να διαβάσει ένα blog για παράδειγμα. Άρα λοιπόν για τους ε, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω είναι προς όφελός τους να δώσουν περισσότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υπολογιστών κτλ. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τους περισσότερους από εμάς είναι πως το διαδίκτυο έχει εκδημοκρατήσει το δικαίωμα της έκφρασης και πως θα πρέπει να έχουμε ένα ίντερνετ με έναν ανοιχτό και ουδέτερο χαρακτήρα. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι μας. Όμως όπως είπαν και οι Κινέζοι φίλοι, αλλά και ο φίλος από το Ιράν, δεν συμβαίνει αυτό παντού. Γιατί τα αυταρχικά ή απολυταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να περιορίσουν τις ελευθερίες αυτές, γιατί με αυτόν τον περιορισμό, αν περιορίσουν τα παραδοσιακά ε, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ε, έντυπος τύπος, ε, τότε πρέπει να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με το διαδίκτυο. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δυτικέ εταιρείε δυστυχώς συνεργάζονται με τα καθεστώτα αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποια θέματα ηθικής, ε, γιατί δυστυχώς στις εμπορικές μας πολιτικές δεν ακολουθούμε πάντα αυτές τις ηθικές επιταγές. Θα μπορούσα να δώσω και κάποια παραδείγματα από πριν από 35 χρόνια, γιατί είναι σημαντικό για την Ευρώπη και για τον μετασοβιετικό χώρο. Τότε είχαμε τη διάσκεψη του Ελσίνκη που έγινε το 1975 και θα θυμόσαστε είχαν τρεις πυλώνες. Είχαμε ε, πολιτική συνεργασία, οικονομική συνεργασία και τρίτος πυλώνας ήταν το κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που βοήθησε να ανοίξουν τα καθεστώτα αυτά και να οργανωθούν κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό μιλάμε και για βραβείο Ζαχάροφ. Η τελική πράξη του Ελσίνκη ήταν όταν η Ελένα Μπόνερ και ο Αντρέι ε, Ζαχάροφ μπόρεσαν να πούνε ότι το έχει υπογράψει η κυβέρνησή μας, το έχει επικυρώσει η κυβέρνησή μας. Άρα λοιπόν αυτά τα δικαιώματα τα θέλουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διδαχθούμε από αυτές τις διαδικασίες όταν αντιμετωπίζουμε καθεστώτα όπως αυτό στην ε, Αφρική που περιγράψατε, στην Κίνα, στο Ιράν, να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ των πολιτικών και στρατηγικών συμφερόντων της οικονομικής συνεργασίας, αλλά και βέβαια ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα άνοιγμα αυτών των κοινωνιών. Αντιμετωπίσουμε όμως και ένα πρόβλημα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι κατά πώς θα πρέπει να επιτρέπεται η νόμιμη παρακολούθηση κάποιας πληροφορίας όταν ε, υπάρχει παραβίαση των ελευθεριών. Για παράδειγμα, με τους παιδεραστές τι κάνουμε. Τι κάνουμε με τους νεοναζί. Τι κάνουμε με ανθρώπους σαν τον Νορβηγό, τον Μπίρβικ. Ε, θα πρέπει να έχουν ανοιχτή πρόσβαση. Θα έπρεπε με τόσο ανοιχτό τρόπο να παραβιάζουν ε, το διαδίκτυο σε βάρος όλων μας ή θα έπρεπε να έχουμε κάποιο τρόπο να παρεμβαίνουμε νόμιμα και να παρακολουθούμε ή να σταματάμε τέτοιου είδους πληροφορίες. Αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το δούμε σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ελευθερία, την ελευθερία της πληροφορίας, την ελεύθερη ροή πληροφοριών αλλά παράλληλα επειδή η δημοκρατία έχει κάποια μέσα για να υπερασπιστεί τον, τις αξίες της, κάτι το οποίο εγώ πιστεύω, γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο ευάλωτοι και τρωτοί που οι δημοκρατίες μας να μπορούν να παραβιαστούν και να χειραγωγηθούν από εγκληματίες, τρομοκράτες, νεοναζί κτλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σε συνεργασία με τους ΜΚΟ μικρών, με τους νομοθέτες, με τους ε, εκπροσώπους των βιομηχανικών κύκλων, να βρούμε ένα κώδικο διοντολογία όπου θα διατηρήσουμε την ελευθερία μεν της πληροφορία την ελεύθερη ροή της πληροφορίας, αλλά παράλληλα θα οικοδομήσουμε και έναν ε, μηχανισμό άμυνας της δημοκρατίας, υπεράσπισης της δημοκρατίας. Δεν λέω πως θα πρέπει να έχουμε λογοκρισία. Δεν θέλουμε λογοκρισία ούτε στον έντυπο τύπο, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο, πουθενά. Ούτε στο ίντερνετ λοιπόν. Αλλά νομίζω που θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συνδυάσουμε την ελεύθερη ροή της προφορίας, την ελευθερία της έκφρασης με την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Λίμπο για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις σα, πολύ χρήσιμε για μας, για τη δουλειά μας, πολύ ενδιαφέρουσες πιστεύω για τους ακτιβιστές, για τους πολιτικούς, για όσους ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα. Και σας ε, παρακαλέσω να είσαστε πίσω στην αίθουσα στις 4 για να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 4 το επόμενο κομμάτι της συζητήσεως. Ευχαριστώ πολύ.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 Yeah. Uh, Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε θερμά σε αυτή τη διάσκεψη. Θα ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση με τους πανελίστες μας. Λέγομαι Edward Macmillan Scott, είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. μάλιστα για πολλά χρόνια ε, ήμουν μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και δημιουργήσαμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό ε, Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την τόσο το τείχους του Βερολίνου. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές και πήγα και επανειλημμένα στην Αίγυπτο πρόσφατα. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα ε, να σας παρουσιάσω τους ε, εισηγητές μας. Όμως να σας πω ότι λείπει, δεν θα είδε εδώ ο Αχμέτ Σαμίχ, ο οποίος ε, είναι ένας νέος Αιγύπτιος ε, διευθυντής του Ινστιτούτου Ανοχής ε, της Ανταλουσίας, ε, μας έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Αίγυπτο αισθάνθηκε υποχρεωμένος να πάει στην Αίγυπτο έτσι ώστε να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο όπου η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά τεταμένη και πραγματικά η σκέψη μας είναι μαζί με τους ανθρώπους που ε, προσπαθούν να συνεχίσουν την ε, επανάσταση στην ε, στην Αίγυπτο και είμαστε σε Είμαστε σε επαφή μέχρι το Σάββατο με την κυρία Καμέλη, η οποία είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια για την Προεδρία, μέχρι το Σάββατο που συνελήφθη ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά ε, και ότι θα φτάσουμε στις εκλογές. Ε, λυπούμαστε. Πάντως ο Αχμέτ Σαμίτ δεν είναι εδώ. Έχουμε μαζί μας τον Σιχέμ Μπεν Σεντρίν, ο οποίος είναι από την Τινησία, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Βαν Ζιαντέχ, ε, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ το Πανεπιστήμιο George Washington. Σιλβάνα Άρμπια, ε, η οποία είναι ε, γραμματέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό τους επόμενους, τις επόμενες εβδομάδες. Κάρλος Βέστεντορπ, Γενικός Γραμματέας της Λέξης Μαδρίτης, παλαιό μέλος του Κοινοβουλίου ε, και ε, διπλωμάτης, ε, Ισπανός διπλωμάτης με μεγάλη Άννα Γκόμες από το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο και Τούνε Κελάμ, ε, μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ασχοληθεί με πάρα πολύ ε, σημαντικά θέματα. Όσον αφορά τώρα τους βραβευμένους, έχουμε την Ασίμα Νασρίνα το 1994, Σαλή Μαχμούντ Μοχάμετ Οσμάνα το 2007 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Δυστυχώς η Λεϊλά Ζάνα δεν θα είναι μαζί μας. Όπως ξέρετε όμως είναι Κούρδος πολιτικός Uh, ε, και ε, ήταν πάντα μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ε, του κουρδικού ζητήματος και που προσπαθούν τώρα να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύμα βίας κατά του κουρδικού λαού. Μούχο Ελίμοβιτς από την Οσλομοντένια ε, πήρε το βραβείο Ζαχάρο το 1993 και βεβαίω ε, θα ακούσουμε παρατηρήσεις και από πλευρά μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω λοιπόν πρώτα τον λόγο με τη σειρά. Δίνω λοιπόν το λόγο στο δεύτερο εγγεγραμμένο, μια και ο Αχμέτ Σαμίχ δεν είναι εδώ, την κυρία Σιχέμ Μπεζρεντίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να εκφράσω την ε, ε, συγκίνησή μου που βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί πραγματικά μου είχατε δώσει επανειλημμένα την ε, δυνατότητα να βρω βήμα για να υπερασπιστώ την χώρα μου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μου. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχής που τώρα μετά από δέκα μήνες ξανά εδώ ενώ η χώρα μου πλέον είναι ελεύθερη και ε, ε, προσπαθεί να οικοδομήσει την δημοκρατία για να πω ότι αυτό είναι δυνατό. Ε, ή να το πω προς τους ανθρώπους που όπως ας πούμε στη Λευκορωσία ε, ε, καταπιέζονται φρικτά και να στραφώ προς αυτούς για να τους πω ότι εάν συνεχίσουμε να τολμούμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία, γιατί η ελευθερία δεν έχει τιμή, τελικά θα καταφέρουν να επιτύχουν την ελευθερία. Πριν από λίγο καιρό ε, είχαμε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Ισία και ο κάθε τιμήσιος άνδρας και γυναίκα ε, αισθάνθηκαν αυτήν την ε, αγαλίαση του να μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους. Η Μισανάβα είναι το πρώτο κόμμα που έλαβε 40% των ψήφων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για, τις, για τα δικαιώματα των γυναικών. Τι σημαίνει αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιος κέρδισε τις εκλογές. Το καλύτερο οχύρωμα ε, για τη δημοκρατία είναι, ε, είναι το σύστημα δικαίου, ε, είναι οι ελεύθερες επικοινωνίες, η ελεύθερη πληροφόρηση, η ελευθερία του λόγου, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να μιλήσει ελεύθερα. Οι τινήσιοι άνδρες και γυναίκες στην ουσία ψήφισαν την ρήξη με το παρελθόν και αυτό πρέπει κανείς να αναγνώσει ως αποτέλεσμα των εκλογών. Ε, ναι, είμαστε μουσουλμάνοι λοιπόν, ναι είμαστε σύγχρονοι, ναι είμαστε ανεκτικοί. Η, το νέο μας ε, κοινοβούλιο, η νέα μας γενική συνέλευση έχει πλέον επιλέξει ε, ως επικεφαλής του έναν ε, δημοκράτη, αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που ε, ήταν ε, πολλά χρόνια αγωνιστής, ο Δόκτωρ Μαζούκη. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε έτσι ώστε να εκπονήσουμε το νέο σύνταγμα, το οποίο θα διασφαλίσει το μήνυμα το οποίο κατέθεσαν οι Τινήσιοι ε, στις ε, τελευταίες ε, εκλογές. Οι πολίτες της Τινησίας κάποια στιγμή σταμάτησαν να φοβούνται. Οι άλλοι άρχισαν να φοβούνται. Άλλαξε στρατόπεδο επομένως, άλλαξε πλευρά ο, φόβος και οι δικτάτορες έφυγαν. Όταν ένας λαός σταματάει να φοβάται, Εκεί ξεκινάει η Επανάσταση σε κάθε χώρα, οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπεραμείνονται της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, θα αλλάξει η κατάσταση. Βεβαίως, πολλή δουλειά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Θα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε, να καθαρίσουμε το σύστημά μας και τη δημοκρατία μας από το φαρμάκι, από το δηλητήριο της δικτατορίας. Να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε ανεκτικοί και ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πιο σοβαρό έργο που έχουμε απέναντί μας είναι βεβαίως το ζήτημα της μεταβατικής δικαιοσύνης ε, εθνική και διεθνής δικαιοσύνη, αποζημίωση των και αποκατάσταση των θυμάτων, προστασία των αρχείων, ε, προστασία των θυμάτων, ε, η δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος για την επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστεί η κοινωνία των πολιτών και οι νέες αρχές ε, ε, οι οποίες ε, τώρα αρχίζουν να κυβερνούν τη χώρα. Αυτό που σας ζητούμε είναι να δείξετε υπομονή, να μην μας ζητήσετε να φτάσουμε στη δημοκρατία κάνοντας ένα μεγάλο άμεσο άλμα. Δεν γίνεται έτσι, ούτε στις χώρες σας έγινε έτσι. Θα πρέπει να δεχτείτε ότι χρειαζόμαστε στη δικιά μας χώρα χρόνο για να μεταβούμε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Να είσαστε λοιπόν κοντά μας έτσι ώστε να μας βοηθήσετε σε αυτή τη μετάβαση. Γιατί ε, σας είπα ότι δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη και ότι είναι εύκολη η μετάβαση αυτή. Πρέπει να πω ότι λίγη πίεση αισθανθήκαμε από πλευρά τη διεθνή κοινότητα προ την παλιά μα κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μπέναλι. αλλά περιμένουμε από τη διεθνή κοινότητα να είναι παραστάτης ε, στην δημοκρατική μετάβασή μας. Πρώτα απ' όλα σεβόμενοι τα αποτελέσματα των ε, πρόσφατων καλπών. Έχουμε εταιρική σχέση μαζί σας ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Ενδεχομένως αυτή η αξιολόγηση γίνεται ήδη από τη δική σας πλευρά. Γιατί κάνοντας την επανάστασή μας εμείς ε, ευνοήσαμε προωθήσαμε και τον τρόπο επαναξιολόγησης αυτής της εταιρικής σχέσης με σας. Ενδεχομένως λοιπόν πολλά ακόμα παραμένουν ε, να γίνουν όσον αφορά την προσέγγιση. Είχαμε πάντα την αίσθηση ότι η Ευρώπη είχε μία προσέγγιση λίγο αφιψηλού και ε, προσπαθούσε να αποτινάξει, ε, να βάλει στο περιθώριο οτιδήποτε ερχόταν από κάτω. Ακόμα και αν ο επίσημος ε, εταίρος ε, είναι σωστός, παρόλα αυτά θα πρέπει κανείς να ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών. Και στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει ε, να ε, ε, ακουστεί η άποψη της κοινωνίας των πολιτών. Εταιρική σχέση δεν είναι μονάχα δεν είναι μονάχα κάποιοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι ξέρουν τα πάντα καλύτερα από μας και θα μας πάρουν από το χέρι να μας γράψουν σχεδόν το σύνταγμά μας. Αυτή την σχέση, αυτή την επαφή δεν τη θέλουμε πλέον. Ο τρόπος με τον οποίο ε, η Ευρώπη υλοποιεί τους μηχανισμούς βοήθειας ή χρηματοδότησης, ε, οι μηχανισμοί στήριξης των μεταρρυθμίσεων, ε, κατά την άποψή μας δεν είναι πλέον διαφανής. Θέλουμε αποσαφηνήσεις, θέλουμε εξηγήσει, θέλουμε διαφάνεια που να τη βλέπουν και τα δικά μας τα μάτια, όχι μόνο τα δικά σας. Από τη δικιά μας πλευρά τα πράγματα δεν είναι σαφή. Αυτή η ίδια Ευρώπη, η οποία συχνά έκανε λάθος απέναντί μας, αυτή η ίδια Ευρώπη, λέγω, έχει δυνατότητες να επανορθώσει τα σφαλματά της. Χρειαζόμαστε αυτή την Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε και μια Ευρώπη η οποία θα μας σέβεται και θα σέβεται τις επιλογές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ροτφαντζιεντή, Σύριος ακτιβιστής που, όπως είπα, μένει στις ΗΠΑ στις 20 Σεπτεμβρίου συνελήφθη ο αδελφός του. Τώρα ευτυχώς έχει αποφυλακιστεί, αλλά τέσσερα ακόμα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται στη φυλακή και γι' αυτό είναι μεγάλη ένδειξη θάρρος το γεγονός ότι έρχεται να μας μιλήσει σήμερα στην ελεύθερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θέλω να πω ότι ιδιαίτερα είμαστε ευγνωμόνε για του ε, αγώνε και τόσο έχετε προσφέρει στα ανθρώπινα δικαιώματα ω Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο και για την ευκαιρία που μα προσφέρετε να μιλήσουμε σε ευρωβουλευτές αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για την κατάσταση στη Συρία. Γνωρίζετε ότι η εξέγερση στη Συρία το Μάρτιο ξεκίνησε μετά την ανατροπή του από την Πεναλή του πρόεδρου της ε, Τινησίας και του πρόεδρου της Αιγύπτου Χωσνή Μουμπάρακ. Ύστερα από εννέα μήνες συνεχών φόνων ε, που χρησιμοποίησε το καθεστώς του Ασάντ εις βάρος του λαού της Συρίας, ο λαός αυτός εξακολουθεί να έχει το θάρρος να κατεβαίνει στους δρόμους και να ζητεί ειρηνικά διαδηλώνοντας το δικαίωμα, το πιο απλό δικαίωμα να αλλάξει πρόεδρο και να μπορεί να επιλέξει την κυβέρνηση που θα τον κυβερνά. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση Ασάντ εξακολουθεί την καταστολή, εξακολουθεί να σκοτώνει τους πολίτες. 32 ήταν αυτοί που έχασαν τη ζωή τους προχτές, μόνο ε- από την πόλη του Χόμς Τη πόλη αυτή που βρίσκεται στο κέντρο τη, Συρία, έξι παιδιά θύματα θρυνήσαμε προχτέ. και 15 σήμερα από ό,τι φαίνεται έκαστον τη ζωή του. Αυτό επιβεβαιώνεται από διαφορετικέ πηγέ. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλλει στην κυβέρνηση, το καθεστώς Ασάτ, να σταματήσει αυτή, αυτή την αιματοχυσία. Είδαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να δράει η διεθνής κοινότητα στο θέμα της ε, Λιβύης. Το ψήφισμα 1970 που καταδίκασε τον Καντάφη, τον Ανουάρελ Καντάφη και που ε, τον παρέπεμπε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάστηκε μόνο έξι μέρες για να εγκριθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Εθνών. Όμως την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ είχαμε επιβεβαιωμένους 3.500 θανάτους στη Συρία και ενώ τώρα ίσως να έχουμε ξεπεράσει και τους 5.000 θανάτους αμάχων πολιτών και όταν έχουμε δύο επιτροπές ανθρωπινών δικαιωμάτων, μία του Απριλίου και μία του Αυγούστου που θέλησαν να επισκεφθούν για να διερευνήσουν ε, εκ μέρους των Εθνών της παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, αλλά απερίφθη αυτό το αίτημα από το καθεστώς Ασάντ, παρότι ζητούσαν απλώς να κοιτάξουν ποια είναι η κατάσταση και ενώ απερίφθηκε το αίτημα πλευρά του Αραβικού Συνδέσμου να αποστείλει παρατηρητέ για την παρακολούθηση τη κατάσταση ε, στη χώρα μα. Ε, μία δε από τι επιφυλάξει προ του παρατηρητέ αυτού από πλευρά του καθεστώτο του Ασάντ είναι ότι δεν θέλουν να του επιτρέψουν να πάνε στα νοσοκομεία διότι ο κάθε ένα από του τραυματίες μα φωνεύτηκε ψυχρό μέσα στα νοσοκομεία. Εάν πάτε να δείτε ε, τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη ζωή τους ε, χωρίς καμία δυνατότητα πρόσβασης στις ε, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο. Αυθαίρετες κρατήσεις επίσης, αυθαίρετες ε, συλλήψεις. Ακυρώθηκε το ποδοσφαιρικό μας πρωτάθλημα διότι ε, όλα, δεσμεύτηκαν μάλλον όλα τα ποδοσφαιρικά μας ε, γήπεδα και κυρίως τις λατάκες της ε, Δαμασκού του Χάμς για να χρησιμοποιηθούν ως στρατόπεδα συγκεντρώσεως ως κέντρα κρατήσεως των πολιτών. Ο αδελφός μου ο ίδιος συνελήφθη τον Αύγουστο, πριν από τέσσερις μέρες μόνο απελευθερώθηκε αλλά ακόμη ένα, δύο μου και τρει από τα ξαδέλφια μου, τον οποίων ο πιο μικρό 14 ετών, βρίσκονται φυλακοί. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει κάτι τέτοιο για μία μόνο οικογένεια. Γι' αυτό έχουμε αριθμού που ξεπερνούν τις 30.000 ε, φυλακισμένων. Γι' αυτό ο καθένας από αυτού του κρατουμένου θα πρέπει και είναι ζωτική σημασία να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην οικογένειά του, σώος και αυλαβή. με βάση διεθνή στοιχεία. Είναι 212 εκείνοι οι οποίοι πέθαναν βασανιζόμενοι στα χέρια των ε, αρχών και υπάρχουν πολλά στοιχεία συγκεκριμένα όπως τη Χάμζα Ελ Χατίμπ 15 ε, ετών και άλλων πολλών που πέθαναν στα χέρια των αρχών στα χέρια της αστυνομίας και του στρατού. Η διεθνή κοινότητα όμως δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένη να κάνει το βήμα αυτό για να βοηθήσει τη Συρία. Και αυτό που ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ακριβώς να αναλάβει δράση. Πριν από δύο ημέρες ή καλύτερα εχθές μόλις ε, η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη ε, συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με 132 ψήφου, δηλαδή 132 κράτη, καταδίκασε τα εγκλήματα του καθεστώτο Ασάντ και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων της, στη Συρία. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι το ψήφισμα τη Γενική Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Πολύ πιο σημαντικό λοιπόν είναι να αναλάβει δράση το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ρωσία, η Κίνα, ξέρουμε ότι έχουν γύρει ζήτημα αρνησικυρίας ως προς το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας πριν από δύο εβδομάδες που μόνο κατά δίκη θα εξέφραζε και δεν θα ζητούσε ε, κυρώσεις τους. Άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα για ε, στρατιωτική επέμβαση. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό που στούμε για τη Συρία και που το συζητούμε εδώ και 10 χρόνια είναι η ανάληψη ευθύνη σε πλευρά τη διεθνού κοινότητα για να προστατέψει του αμάχου. Είναι σαφέ ότι δεν θα σταματήσει αυτούς του, αυτή την αιματοχυσία το καθεστώ του Ασάντ. Κάθε μέρα κατεβαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο, κάθε μέρα αντιμετωπίζουν ε, του ε, ένοπλους, της πολιτοφυλακές του καθεστώτος, τους παραστατικούς μάλλον του καθεστώτος ε, και τους ε, φόνους αυτούς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσει η Εθνική κοινότητα. Αν μπορέσει να δείξει αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση αυτών των, ε, αυτής της καταστολής και σε τελευταία ανάλυση πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει σε τίποτα αλλάξει το καθεστώς η εξέγερση της, στη Συρία χαρακτήρα παραμένει μια φιλιρινική ε, εξέγερση ενώ το καθεστώ χρησιμοποιεί ακόμα και αεροπλάνα για να βομβαρδίσει του Αμάχου. Αυτό που ζητούμε λοιπόν τώρα είναι να λάβει αποφασιστικά δράση εθνή κοινότητα για να προστατεύσει του Αμάχου, για να εξασφαλίσει μια ουδέτερη ζώνη στα σύνορα με την Τουρκία, για να εξασφαλίσει την απαγόρευση των υπερπτήσεων, για να αποτρέψει του βομβαρδισμού. Τα σύνορα με την Τουρκία θα μα επιτρέψουν να έχουμε ένα ασφαλή χώρο διαφυγής και ταυτόχρονα θα μπορούν να εξετάσουν την κατάσταση και διεθνεί παρατηρητέ όπω έγινε το 1995 στο Κοσμοπέδιο όπου τα Ηνωμένα Έθνη απέστειλαν 7.000 παρατηρητέ και ανώκρανου για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να καταγράψουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά του Συμβουλίου Ασφαλεία για να αναλυφθεί δράση. Αλλά δυστυχώ ακόμη δεν έχουν αναλυθεί τα μέτρα αυτά που χρειάζονται τόσο αδέρυτα για την προστασία των αμάχων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω τώρα στην ε, Σιλβάνα Άρβια που είναι νομικός, έγινε γνωστή ε, στο Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και είναι αυτή τη στιγμή και γραμματέας του Διεθνής Δικαστηρίου στη Χάγη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Στα γρήγορα να σας πω πως εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσκληση αυτή να έρθω σε αυτή τη συνεδρία όπου θα συζητήσουμε αυτή την πρόθεση της ε, δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προέρχομαι από οργάνωση του Διεθνές Ποινικού Δικαστήριο που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών είτε πρόκειται για κατηγορούμενο ή ύποπτο, είτε πρόκειται για ε, θύμα ή μάρτυρα που χρειάζεται προστασία ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με τους ιδιώτες, με τα άτομα και προσπαθούμε να προσφέρουμε τα, τις βέλτιστες προδιαγραφές προστασίας, τις βέλτιστες ε, προδιαγραφές ε, ισότιμης δίκης. Ένα φιλόδοξο σχέδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλλει σε αυτό, καθώς ε, έχουν ε, προσυπογράψει τη συνθήκη, το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τα 27 κράτη-μέλη και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι ξεκάθαρο από το καταστατικό ότι ο στόχος ε, των ιδρυτικών κρατών, των κρατών μερών, είναι αυτός ακριβώς. Έχουμε μεταξύ 119 κράτη-μέρη στο καταστατικό της Ρώμης. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι κοινή οι δεσμοί, είναι κοινή η κληρονομιά των λαών και κοινή η ανησυχία μην ανατραπεί αυτό το μοσαϊκό των αξιών που είναι τόσο ευάλωτο. Γι' αυτό θεσπίστηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ιδρύθηκε λοιπόν και ως καθήκον των κρατών να ασκήσουν την ποινική τους δικαιοδοσία ε, εις βάρονες εκείνων που έχουν την ευθύνη διάπραξης διεθνών εγκλημάτων. Η ατιμορρησία λοιπόν ήταν ο κύριος στόχος της, ε, της διεθνούς κοινότητας. Η ατιμορρησία που μπορούμε να καταπολεμήσουμε με το μέσον αυτό της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης που είναι έτοιμη να παρέμβει σε κάθε σχετική κατάσταση και έχει τους μηχανισμούς έθεση για να επιβάλλει την, ε, ε, το δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ε, τις τελευταίες μέρες με την σύλληψη του Απτούλ Σαμούση και του Σαΐφ Αλισλάμ Καντάφη, τους δύο αυτούς που συνελήφθησαν στην ε, ε, Λιβύη και για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για κατηγορίες διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι η Λιβύη είναι συμβαλόμενο μέρο στο καταστατικό mm. της Ρώμης, που θεσπίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είχε την υποχρέωση να, είχε την υποχρέωση να συλλάβει και να ε, παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τους δύο αυτούς υπόπτους. Τι είναι λοιπόν το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο σήμερα, γιατί σήμερα και ποιο είναι ο κεντρικό μα ρόλο μεταξύ άλλων νομοθετημάτων και μέσων προστασία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί μια πραγματικότητα, αποτελεί ε, ένα δικαστήριο που αντιμετωπίζει ε, πτά διαφορετικές καταστάσεις, ασκεί δικαιοδοσία ως προς διεθνή, ε, σοβαρότατα διεθνή εγκλήματα σε 7 διαφορετικά κράτη δηλαδή. και είτε πρόκειται και μια πολιτική απόφαση, δηλαδή την παραπομπή από ένα κράτο ε, μια υπόθεση στο δικαστήριο, όπω έγινε με την, ε, Ρουάντα, με την τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ή την παραπομπή από ένα συμβούλιο, από το Συμβούλιο Ασφαλεία, όπω έγινε με την περίπτωση του Σουδάν, του Νταρφούρ συγκεκριμένα, είτε πρόκειται για την παραπομπή ή την προσφυγή καλύτερα ενό κράτους μέρους η εισαγγελία του Εθνικού Ποινικού Δικαστηρίου μπορεί να ξεκινήσει και πέραν αυτών των δυνατοτήτων και δική τη ε, έρευνα. Πρόκειται δηλαδή για ένα ε, μέτρο πάρα πολύ σημαντικό, ένα μέσον πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να εξασφαλίσει ισότιμα, ε, ισότιμες προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας των θυμάτων. Έχουμε πάνω από 9.000 θύματα τα οποία έχουν, ε, έχουν υποβάλει έτσι για συμμετοχή στις διαδικασίες του δικαστηρίου. Πέραν των αριθμών, ε, η σημασία έχει το τι προσδοκούν αυτά τα θύματα. Τα θύματα αυτά προσδοκούν αποκατάσταση, αποζημίωση. Επομένω, οι δύο πολύ σημαντικέ έννοιε, οι δύο σημαντικοί πυλώνες πάνω στους οποίου χτίζεται η υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Δικαστήριο είναι το, η πέραση της και η αποκατάσταση για τα θύματα. Πέραν αυτού όμω, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο εξαρτάται από τη συνεργασία των ε, κρατών, από τη συνεργασία των διεθνών οργανισμών και οργανώσεων, από την υποστήριξη τη της κοινωνίας των πολιτών και ακριβώ αυτό ε, προλαμβάνουμε διαρκώ αυτό υποστηρίζουμε ε, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το δικαστήριο είτε να συλλάβει είτε να παγώσει περιουσιακά στοιχεία είτε να επιβάλλει αποκατάσταση. Είναι απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία των κρατών μερών, είναι πολύ σημαντική η πολιτική τους υποστήριξη όπως εκφράζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιο συγκεκριμένα, το οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερω για την ερετή υποστήριξη που προσφέρει στα ψηφίσματά του, αλλά και ιδιαίτερα και τους λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η σημασία όμως ξέρετε ότι έχει και ο προπολογισμό του δικαστηρίου, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι παρά την αύξηση του φόρτου εργασίας και των δραστηριοτήτων του δικαστηρίου που δραστηριοποιείται, όπως είπα σήμερα, σε 7 χώρες και προσπαθεί να εξασφαλίσει ισότιμο πεδίο προδιαγραφών και από προστασία και ε, στήριξη προς τα θύματα στις 7 αυτές χώρες πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ε, Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Δηλαδή υποστηρίζουν μηδενική αύξηση στον προπολογισμό. Και ενώ αναγνωρίζεται η σημασία αυτού του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου και η τελευταία μάλιστα παραπομπή τη Λιβύη ε, ε, από πλευρά του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι πιστεύω η σεφέστερη απόδειξη ότι συμβάλλει στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο ε, Δυστυχώ κάποια κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να εξασφαλίσουν και του απαραίτητου πόρου που χρειάζεται το δικαστήριο για να κάνει ακριβώ αυτό που είναι απαραίτητο να πράττει, δηλαδή να λειτουργεί, να εκδικάζει, να ασκεί την εντολή του όπω οφείλει. Αυτό είναι ένα κύριο πρόβλημα και ε, η απουσία μερικών εκατομμυρίων ευρώ μπορούν να αποτελέσει το λόγο μπορεί να παρεμποδίσει την ουσιαστική αποτελεσματικότητα των εργασιών του δικαστηρίου μας. Μια εμπειρία λοιπόν γνωστή, μεγάλη εμπειρία, υπηρεσία πολύ σοβαρή που μπορεί να προσφέρει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην ανθρωπότητα κινδυνεύει για μερικά εκατομμύρια ευρώ δεν είναι κάτι το ίσονο σημασίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το θέμα του προϋπολογισμού. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη των κρατών μελών, χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη τους. Αυτή σημαίνει όχι μόνο ηθική ε, υποστήριξη, αλλά και υλική, πραγματική υποστήριξη. Και χρειαζόμαστε τους πόρους για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Πέρας λοιπόν ε, της ε, ατιμορρησίας ένα εγχείρημα το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Ε, η ανθρώπινη δραστηριότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδια σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ισχύουν κάπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν, υπάρχουν, δεν ισχύουν κάπου αλλού. Αυτό ακριβώς βρίσκεται και στο επίκεντρο του σχεδίου για το πέρας της ατιμορρησίας. Εγώ έρχομαι από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα γιατί και είμαι υπερήφανη για την ε, ανάπτυξη και λειτουργία του. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, να, προσφέρει, να προστατέψει τους, τα θύματα, να προσφέρει δηλαδή στήριξη στα θύματα και μετά από πολύ ε, τραγικές εμπειρίες. Από την άλλη όμως φοβούμε ότι κινδυνεύει το εγχείρημα αυτό κινδυνεύει, αλλά δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να ανατραπεί. Χρειάζεται η στράτευση και υποστήριξη των κρατών μερών και γι' αυτό ελπίζω ότι θα πάτε όλοι τον Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω ότι θα δούμε την υποστήριξη των κρατών μερών, των κρατών σας και ελπίζουμε ότι τα 27 κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρη συμβαλόμενα του καταστατικού της Ρώμης, ε, όχι όμως μόνο αυτά, θα δώσουν την υποστήριξη της. Γιατί πέραν αυτών των 27 χρειαζόμαστε την υποστήριξη των λοιπών κρατών μερών, χρειαζόμαστε τη στήριξη της ε, κοινωνίας των πολιτών, χρειαζόμαστε την εδραίωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και την εμπιστοσύνη στη δουλειά του. Υπάρχουν πολλά θέματα. Με την ε, ε, πιθανή καταδίκη του Λουμπάγκα θα μπορέσουμε πιστεύω να φτάσουμε στη συζήτηση της αποκατάστασης για τα θύματα και άρα θα έχουμε την πρώτη ουσιαστική δράση του δικαστηρίου υπέρ των θυμάτων με την αποκατάσταση. Εκεί θα δούμε πραγματικά πόσο σημαντικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα έπρεπε να έχω κάνει μια εισαγωγή και να παρουσιάσω και την Μπάρβαρα Λόκπιλα, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα κάνει κάποια ε, τελικά σχόλια. Ο Κάρλος Βέστεντορπ, και δεν θα πειράξει, δεν τον πειράξει που το λέω, είναι βετεράνος διπλωμάτης και ήταν ε, και αρμόδιος ε, για τις διαπραγματεύσεις που έφεραν την Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι χαίρονται που είναι μέλη σήμερα. Είναι λοιπόν από το κλαπ της Μαδρίτης και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με επιτρέπει να ε, γυρίσω ε, στο χώρο αυτό και για να τονίσω τη σημασία που έχει η στήριξη δημοκρατίας στις μεταβατικές αυτές ε, περιόδους. Και θα ήθελα να πω σε όλους όσους μάχονται υπέρ της δημοκρατίας, οπουδήποτε και να βρίσκονται, και κυρίως να πω σε όσους έχουν βραβευθεί με τα βραβεία Ζαχάρ, πως χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχετε θέσει επιτάπητο στο θέμα της πολιτικής ηγεσία και του διαλόγου που είναι σημαντικά και είναι ακόμα πιο σημαντικά όταν σκιάζονται από άλλες προτεραιότητες. Όταν δεν τα εκτιμούν αρκετά και όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ε, οικονομικών συμφερόντων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώς πολύ συχνά τα οικονομικά συμφέροντα επιβάλλονται. Στο τέλος, όπως είχε πει και ο Βάτσλαβ Χάβελ, το κόστος είναι πολύ ψηλό. Το αντίτιμο είναι πολύ υψηλό και τελικά ξεπερνά και τα ίδια τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία επιδιώκαμε. Ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από την εμπειρία που έχω από τις προηγούμενες μου θέσεις και στην κυβέρνηση αλλά και σε άλλα σημεία είναι το εξής. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε εγχειρίδιο για το πώς να ηγηθεί κανείς μιας μετάβασης προς τη δημοκρατία. Πρόεδροι, ηγέτες, πρωθυπουργοί σε χώρες που γέννησαν τέτοιες μεταβατικές περιόδους προς τη δημοκρατία ε, έκαναν προσπάθειες για να οικοδομήσουν θεσμούς δημοκρατικούς ε, και φορείς δημοκρατικούς ε, χωρίς να έχουν τέτοιο είδος εγχειρίδιο να τους βοηθήσει. Πολλές φορές όμως ζητούν στήριξη από το εξωτερικό. Θέλουν να ενημερωθούν για το ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, χρειάζονται πολιτική καθοδήγηση και ε, στρατηγικές συμβουλές. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Κλαμπ της Μαδρίτης που μπορεί να το καταφέρει γιατί αποτελούμαστε από 87 πρώην ε, αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών από πάνω από 60 κράτη οι οποίοι διαθέτουν χρόνο, εμπειρία για να προωθήσουν τη δημοκρατία παντού. Όλοι παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα κύματα αυτά κινημάτων λαών που ζητούν περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Και μάλιστα με την ανάφλεξη στην την Ισία πέρυσι και τη διάδοση στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούμε πως ε, αποτελεί ένα ε, φάρο ελπίδας και με πολύ ενθουσιασμό ε, αυτή η ελπίδα για ευημερία και δημοκρατία έχει ριζώσει στις χώρες αυτές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι τεράστιες. Αλλά η... το καθήκον του να οικοδομήσει δημοκρασία, τη δημοκρατία ποτέ δεν τελειώνει. Γιατί καμία δημοκρατία δεν είναι τέλεια και καμία δεν είναι πλήρης. Η εγκαθίδρυσή της χρειάζεται χρόνο και στις μεταβατικές φάσεις και όταν η ορίμανση είναι χαμηλή παρουσιάζονται κάποιες ευκαιρίες αλλά και εξαφανίζονται με την ίδια ταχύτητα με την οποία εμφανίστηκαν. Και στην στιγμή αυτή οι μεταρρυθμιστές χρειάζονται τη δική μας εξωτερική στήριξη. Η εμπειρία που έχουμε ως μέλη του κλαμπ της Μαδρίτης, γιατί πολλοί από εμά έχουμε ε, συνδεθεί με την δημοκρατική μετάβαση των χωρών τους, ε, μας προσφέρουν ε, τα όπλα για να βοηθήσουμε ε, ο Ρικάρος Λαγός στη Χιλία, ο Φελίπο Γκονζάλες στην Ισπανία, ο Βάσιλαβ Χάβελ στην Τσεχία, ο Μουγέτης της Αγκόλα. Κάθε μετάβαση είναι διαφορετική και η πολιτική δράση που χρειάζεται είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζουμε όμως ότι να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές συνέπειες αυτής της μετάβασης είναι μία μακρά διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας αποτελεί τον κατάλληλο διεθνή παίκτη που θα στηρίξει αυτή τη διαδικασία τις πρώτες μέρες μετά την εκκίνηση της μετάβασης προς την δημοκρατία. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις εμπειρίες που είχαμε. Αϊτή, Κυργιστάν και Τιμόρ Λέστε. Στις τρεις αυτές προσπάθειες που κάναμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας βοήθησε να ε, συμβουλέψουμε αυτούς τους ηγέτες και να τους δώσουμε κάποια στοιχεία για να πάρουν αποφάσεις στις κατάλληλες στιγμές. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Η δημοκρατία έχει προχωρήσει χωρίς βεβαίως να έχει παγιωθεί. Θα ήθελα να επιστρέψω στην εισαγωγή που έκανα. Το κίνημα της Αραβικής Άνοιξης το παρακολουθεί ολόκληρος ο κόσμος με θαυμασμό και με ελπίδα και κυρίως οι νέες γενιές ε, εξασφάλισαν πως ακούστηκαν οι φωνές τους και αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό για την αλλαγή. Δικαιοσύνη, ελευθερία ήταν ε, τα συνθήματά τους και έχουν φέρει συνδίκες ανεξαρτησίας για πάρα πολύ κόσμο, δημιουργώντας καινούριε προσδοκίες στις χώρες αυτές. Ο θαυμασμός και η ελπίδα δεν θα πρέπει όμως να μας τυφλώνουν για τις τεράστιες προκλήσεις που έχει το μονοπάτι για την ευημερία, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία. Σε όλη την περιοχή αυτή η οικονομική κατάσταση είναι ασταθής και υπάρχει αυτός κίνδυνος αυτό να παρακολύσει, να παραμορφώσει και τις διεθνείς αλλά και τις εθνικές ελπίδες για μια πιο σταθερή ε, και ευκολή μετάβαση. Είναι καθήκον μας να τους βοηθήσουμε, αλλά μας συμφέρει κιόλα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά συμφέροντα, ευτυχώς στην περίπτωση αυτή, ε, συνοδεύουν ε, το ένα το άλλο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλο το πάνελ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όσους έχουν βραβευθεί Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ναζρίν που είναι συγγραφέας από τον Μπαγκλαντές να μας κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι πιστεύουμε πως η δημοκρατία είναι καλύτερη από τη δικτατορία. Ακόμα και μια διεφθαρμένη δημοκρατία. Ακόμα και αν οι ηγέτες μας δεν είναι κατάλληλοι και θέλουμε να τους διώξουμε. Η δημοκρατία και πάλι είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία όταν δεν ακούγονται οι φωνές των γυναικών. Πιστεύω ότι το 50% των γυναικών, μάλλον στο κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχουμε κοροσώπηση 50% από γυναίκες. και πως υπάρχει μια συνωμοσία η οποία αποκλεί τις γυναίκες από την πολιτική. Άντρες με πατριαρχικά και θρησκευτικά και παραδοσιακά πολιτιστικά πρότυπα δεν θέλουν οι γυναίκες να έχουν κυβερνητικό ρόλο. Δεν μπορούμε να πετύχουμε πραγματική δημοκρατία εάν δεν υπάρχει χωρισμός εκκλησίας και κράτους, χωρισμός της εκκλησίας από το δικαστικό και εκπαιδευτικό σύστημα. Not with Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα γυναικεία δικαιώματα και η δημοκρατία, ο λαϊκισμός, η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορούν να συνδυάζονται με ε, θρησκευτικά καθεστώτα. Το πρόβλημα είναι πως ο κόσμος είναι θρησκευόμενος. Και πολλές φορές δεν επιθυμούν κοσμικό κράτος γιατί έχουν υποστεί ε, μια προπαγάνδα από τους φουνταμενταλιστές, τους θρησκευτικού φουνταμενταλιστές, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν μια θεοκρατία. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στους φανατικούς αυτούς να καταστρέψουν τις δημοκρατίες μας και τις αρχές τις δημοκρατικές που ισχύουν. Τα άτομα αυτά τα οποία προωθούν ε, τον Ισλαμικό νόμο, τη Σαρία, που κάνει διακρίσεις εναντίον των γυναικών, πετροβολούν γυναίκες, φοράνε μπούρκα στις γυναίκες και τις υποχρεώνουν να ζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ως απλές μηχανές που γεννάνε παιδιά, αντικείμενα σεξουαλικής υποδούλωσης. Η κοινωνία των πολιτών αποτελείται από ανθρώπους με τελείως διαφορετικές ιδέες και πιστεύω. Και νομίζω ότι οι καλύτερες από αυτές θα έπρεπε να χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης άνθρωποι, γυναίκες και άντρες με κοσμικές ε, πεπιθήσεις θα πρέπει να έχουν ηγετικέ θέσεις και δεν θα πρέπει να αφήσουμε την ηγεσία μας ε, στις γυναίκες που φορούν μπόρκα και σε αυτόν που τους επιβάλλουν να τη φορέσουν και που προσπαθούν να επιβάλλουν αυτά τα ε, συστήματα, τα πατριαρχικά, τα παραδοσιακά, τα φανατικά ε, δεν θα έπρεπε να του επιτρέψουμε να είναι οι, οι μελλοντικοί μας ηγέτε. Η θρησκεία θα πρέπει να μένει στον προσωπικό χώρο και όχι στο δημόσιο χώρο. Και δεν μπορεί να συνδυαστεί η θρησκεία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα γυναικεία δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και τις δημοκρατικές αρχές. Δεν πιστεύω πως οι γυναίκες αν λάβουν κυβερνητική θέση θα λύσουν όλα τα προβλήματα των γυναικών στη χώρα τους. Στη δική μου χώρα, τον Μπαγκλατές, είχαμε πρωθυπουργό γυναίκα, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης γυναίκα για δεκαετίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία ιδεολογική δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της θέσης των γυναικών στη χώρα μου. Στην ε, Ινδική ε, Χερσόνησο και ε, στη χώρα μου ε, σκοτώνουν τα κορίτσια όταν γεννηθούν. Υπάρχει εμπορία γυναικών, σεξουαλική υποδούλωση, εκπόρνευση, ε, φόνη για την πρίκα, ε, βιασμοί, ομαδικοί βιασμοί, σεξουαλική παρενόχληση. Αυτά έχουν υποστεί οι γυναίκες στη χώρα μας και οι χώρες μας θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες για τη γυναίκα στον κόσμο. Παρόλο που πολλές φορές φτάνουν σε θέσεις εξουσίας οι γυναίκες. Δεν κάνουν οτιδήποτε για να βελτιώσουν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας. Γιατί δεν έχει σημασία το φύλλο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ιδεολογική δέσμευση για την βελτίωση της θέσης των γυναικών που είναι σημαντική. Αυτές οι δύο γυναίκες χρησιμοποίησαν τη θρησκεία για να τις ψηφίσουν οι αμόρφωτες μάζες. Δεν με αφήνω να γυρίσω στη χώρα μου γιατί έγραψα βιβλία για τα δικαιώματα των γυναικών που έρχονται σε αντίφαση με τους Ισλαμικούς νόμους. 17 χρόνια ζω εξόριστη. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να έχουμε κοσμικό κράτος με μη θρησκευτικούς εκπροσώπους, άντρες ή γυναίκες στην εξουσία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εκκοσμικευθούν τα Ισλαμικά συστήματα, οι νόμοι και τα και το εκπαιδευτικό σύστημα και να υπάρχει πραγματική διάκριση και διαχωρισμός μεταξύ, ε, θρησκείας και κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Σαλή Οσμάν ε, από το Σουδάν ο οποίος ε, έδωσε δωρεάν την νομική του ε, βοήθεια σε πολλούς κατατραγμένους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων που μου δίνετε για μία ακόμα φορά ε, στα πλαίσια της βράβευσής μας με το γραφείο Ζαχάροφ που μας δίνετε λέω τη δυνατότητα να ξαναέρθουμε εδώ για να μιλήσουμε ε, για αυτά τα σημαντικά θέματα. Θα ήθελα απευθείας να, να ασχοληθώ ε, με, τον, ε, με, το θέμα μου, δηλαδή τη μετάβαση προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν. Μετά το τέλος του CPA βεβαίως έπρεπε να προχωρήσουμε στη μετάβαση προς τη δημοκρατία. πολλές υποσχέσεις είχαμε ακούσει όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη νέα διακυβέρνηση και τη δημοκρατία στις, ε, στη χώρα μου. Δυστυχώς όμως ε, είχαμε εκλογές οι οποίες δεν έγιναν με σωστό τρόπο. Οι παρατηρητές από άλλες χώρες είπαν απλώς ότι αναφέρθηκαν κάποιες ε, ανομαλίες και ότι τέτοιου είδους ανομαλίες ε, είναι συχνές ε, στις αφρικανικές χώρες. Εμείς όμως, για μας αυτό είναι προσβολή. πρέπει να έχουμε ίδια δικαιώματα με τα άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας και όταν υπάρχουν ανομαλίες που καταγράφονται από τη διεθνή κοινότητα, τότε, τότε η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να μπορεί να πει ότι δεν είναι το να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Δυστυχώς όμως δεν έγινε έτσι. Αποτυχία λοιπόν σε κάθε επίπεδο και όσον αφορά το αποτέλεσμα, σαφέστατα δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση του κόσμου. Ξέρω πάρα πολύ καλά, σαν δικηγόρος, ότι ήταν δικαίωμα των, ε, των κατοίκων του Νότου να ζήσουν ελεύθερα και να μην έχουν πλέον αυτό το καθεστώς καταπίεσης. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έγιναν τα πράγματα δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Όταν ε, μιλάμε λοιπόν για μετάβαση προς τη δημοκρατία, χρειάζονται κάποιες ε, συγκριτικές αξιολογήσεις, ε, ας πούμε. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη για τις καταστάσεις στον Ταρφούρ και στις νότιες περιοχές της χώρας, τότε αυτό ο πόλεμος, ο οποίος τελικά κατέληξε σε γενοκτονία, σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, θα έπρεπε ε, να είχε αντιμετωπιστεί καλύτερα ε, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου της, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα έπρεπε να είχαν φτάσει όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι για τον Ταρφούρ. Όμως δυστυχώς καμία δράση δεν ανελήφθη από τη διεθνή κοινότητα, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι των φρικτών αυτών πράξεων να φτάσουν ε, ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκατοντάδες ε, ήταν οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων, των παραβιάσεων ε, που χαίρουν ατιμορρησίας, δεν, δεν τους αγγίζει η δικαιοσύνη. Ε, στην ε, ε, νότια, στο νότιο τμήμα της χώρας τα πράγματα εξακολουθούν να είναι και πάρα πολύ δύσκολα, αλλά βεβαίως όχι μόνο σε εμάς και στην Αίγυπτο και στην Ινσία, στην Λιβύη τούτη τη στιγμή που μιλάμε, στη Συρία. Όλοι βλέπουμε καθημερινά να χάνονται ανθρώπινες ζωές και κανείς ε, δεν ε, αναλαμβάνει δράση έτσι ώστε να σταματήσει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για δημοκρατία όταν η διεθνής ε, κοινότητα έχει κατά νου μονάχα τους συμβιβασμούς. Στην Αφρική έχουμε υποφέρει πολύ από αυτό. Χρειαζόμαστε μια ε, ενωμένη αντικατάσταση, ε, ε συγγνώμη, μια οργανωμένη ε, εκπροσώπηση και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται λόγος πλέον για τη Συρία και για το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι ε, πρωταρχικό μέλημα. Να τελειώσω λέγοντας δύο λόγια για τη χώρα μου, για το Σουδάν. Πρέπει ενεργά να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα όλων των ε, ε, πολιτών του Σουδάν, γιατί είμαστε μια πολυφιλετική κοινωνία. η παρούσα κυβέρνηση εξακολουθεί την ίδια ε, ε, πολιτική της καταπίεσης των πληθυσμών του Νότου και συγκαταλέγει στους φανατικούς οποιονδήποτε προσπαθεί να ορθώσει το ανάστημά του. Νομίζω ότι η ε, διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει δράση έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τον κύριο Σιλέμοβιτ από την εφημερίδα της Βοσνίας Αρζογοβίνης. Κυρίες και κύριοι, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ το θέμα του τι έγινε από τότε που δώσαμε το βραβείο μέχρι σήμερα, γιατί από τότε που το πήρα πέρασαν 18 χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς δράσαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της ισοστορία μας, στην περίοδο του πολέμου όπου προσπαθούσαμε κάθε μέρα να τυπώσουμε την εφημερίδα μας για να τηρήσουμε ενήμερο το κοινό μας. Ε, τους αναγνώστες μας. Μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα μου. Όπως είπα, οι δημοσιογράφοι μας ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης και προσπαθούσαν να κρατηθούν ζωντανοί. Όταν λοιπόν μας δώσατε το βραβείο, το κτίριο στο οποίο δουλεύαμε βομβαρδίστηκε. Καταστράφηκε πλήρως. Και με αυτό έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Όσο άσχημη και να είναι η κατάσταση μέσα στην οποία ζει κανεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπνίξει κανείς αυτούς οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τις αρχές οι οποίες όλος πιστεύουμε. Η Ασλαβατζένια έγινε το σύμβολο ε, της βοσνιακής κοινωνίας. Εκείνη την εποχή ζούσαμε μέσα σε ένα πόλεμο και είχαμε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά συμφέροντα, κροατικά, σερβικά, βοσνιακά. Εμείς γεννηθήκαμε για να γίνουμε μια εφημερίδα που θα προωθούσε την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατία, ε, δικαιώματα τα οποία έχουμε εδώ και χρόνια κατακτήσει στη Βοσνία. Αλλά ε, πρέπει να σας πω πως ε, όταν έγινε ο πόλεμος τα δικαιώματα αυτά κατέρευσαν και εμείς ήμασταν πάντα ανοιχτοί για όλους στη Βοσνία, για τους Κροάτες, για τους Μουσουλμάνους, για τους Σέρβους και ίσως αυτό για εσά του Ευρωπαίου να φαίνεται φυσιολογικό. Αλλά αν ξέρατε πόσο περίπλοκη είναι η κοινωνία μα, θα ξέρατε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Δώσαμε τεράστιε μάχε για να έχουμε αυτή την ισότιμη εκπροσώπηση. Στη χώρα μα δώσαμε τη μάχη για να κατακτήσουμε κάτι το οποίο εσεί στη χώρα σα θεωρείτε φυσιολογικό. Η ασλαμπαζένια, που σημαίνει απελευθέρωση, είναι ένα, α, μια εφημερίδα που περιγράφει τα εγκλήματα όποιος και να τα έχει διαπράξει. Και όταν μας δώσατε πριν από 18 χρόνια το βραβείο, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα. Σήμερα στη Βοσνία πολλά έχουν βελτιωθεί. Και αληθεύει πως τα δικαιώματα για τα οποία οι Βόσνοι πολεμήσαμε, στην πλειοψηφία τους έχουν παγιωθεί. Για παράδειγμα, ε, στην ιδιωτική περιουσία, στο να είναι κανείς διαφορετικός, στη ζωή, στην ελευθερία ε, του να επιλέξει κανείς την φυλετική του ταυτότητα. Εμείς δώσαμε τη μάχη στα ΜΜΕ και ήμασταν πάντα σε επαφή με τους εκπροσώπους των διαφορών πολιτικών ομάδων στη χώρα μας. Πολλοί από εμάς μάλιστα πέσαμε και θύματα του εθνικισμού. Όμως αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει στη χώρα μας είναι το εξή. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό ακόμα είναι απαραίτητο να αγωνιζόμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω τώρα να δώσω την εντύπωση πως τα δικαιώματα τα οποία όντως παγιώσαμε ε, είναι δικαιώματα τα οποία θεωρούμε αυτονόητα. Όχι, γιατί έχουμε κάποια άλλα δικαιώματα που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Υπάρχει ακόμα μίσος στην καθημερινότητά μας. Βασίζεται σε κάποιες διαφορές περιφερειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, φιλετικές και θα πρέπει να συνεχίσουμε στηρίζοντας το δικαίωμα που έχουμε καταρχήν στην ιδιοκτησία και όσοι χρειάστηκε να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα χέρια τους στον πόλεμο να μπορούν να επιστρέψουν και να τους επιστραφούν οι περιουσίες τους. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ε, με την ανεργία. Πάνω από το 40% του πληθυσμού δεν έχει δουλειά. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε και τη μάχη για μια αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα η μάχη που δίνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται με δυσκολίες. Αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε εναντίον στοιχείων που χρησιμοποιούν όλο και πιο προχωρημένους τρόπους για να μας καταπολεμήσουν εμάς τους ακτιβιστές που προωθούμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Κάθε φορά είναι όλο και πιο ε, προχωρημένα τα μέσα που βρίσκουν για να, μας, για να πνίξουν τη φωνή μας. Εμείς δίνουμε τη μάχη κατά, ε, κατά των εξτρεμιστών, της εγκληματικότητας, ε, της διαφθοράς, όπου και να βρίσκεται στη βοσνιακή κοινωνία. Και από τότε που μας δώσατε το βραβείο, ε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί το βραβείο Ζαχάροφ στηρίζει ομάδες που προωθούν τα δικαιώματα αυτά. Είμαστε από μια μικρή χώρα και πολλές φορές η μάχη που δίνουμε υπέρ της δικαιοσύνης και υπέρ ε, του καλού είναι ε, μια μάχη στην οποία αισθανόμαστε απομονωμένοι, ασήμαντοι πως οι υπόλοιποι δεν αναγνωρίζουν το έργο μας, δεν γνωρίζουν τι κάνουμε καν. Γι' αυτό υπάρχουν ακτιβιστές οι οποίοι έχουν καλές προθέσεις, αλλά επειδή δεν στηρίζονται, τελικά τα παρατάνε. Εγκαταλείπουν την προσπάθεια και εγώ τους λέω, αξίζει τον κόπο να δώσεις τη μάχη για αυτό που είναι δίκαιο και σωστό. Και νομίζω ότι αυτό μαρτυρούν και οι, ε, οι καλεσμένοι σήμερα. Δεν λύγησαν μπροστά στα εμπόδια. Απέδειξαν πως αξίζει τον κόπο να αγωνιστείς, γιατί ο αγώνας αυτός θα δώσει καρπούς. Και στον κόσμο μας ακούνε. Υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί, που μας στηρίζει. Ξέρει τον αγώνα μας και είναι δυνατόν να κερδίσεις. Καμιά φορά καθυστερεί η νίκη, αλλά δεν χρειάζεται κανείς να εγκαταλείπει τη μάχη. Και εμείς θέλουμε μια Βοσνία η οποία θα είναι μια κοινωνία ενωμένη, παρόλο που είναι πολύ περίπλοκη, με πολλά προβλήματα, αλλά θα δώσουμε τη μάχη για την αλήθεια, για την δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Ε, και τώρα, όπως είπα, νωρίτερα η Ρέλα Ζώνα δεν μπόρεσε να έρθει στις Φρυξέλλες, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιος βρίσκεται εδώ για να διαβάσει το μήνυμά της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Το μήνυμα της Ζάνα είναι στα τουρκικά και πριν το διαβάσω θα ήθελα να παρουσιάσω, να υποβάλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της Τενέλη Μητεβαγών που ήταν γνωστή και ως μεγάλη πρόσπιση των δικαιωμάτων και των Κούρδων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι ε, βραβευτέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να εκφράσω να μας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μου δίνετε να βρισκώ εδώ. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν θα ήθελα να πω ότι άκουσα την είδηση για τη θέσπιση αυτού του δικτύου ε, Ζαχάροφ. Με πολύ μεγάλη χαρά ε, έρχομαι, μαθαίνω μάλλον την είδηση για την εγγενείας και μία αίθουσα που φέρει το όνομα του Ζαχάροφ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και παραβιάσεις ανθρώπων δικαιωμάτων και δεν είναι δυνατόν να τα απαριθμίσω όλα. Ήταν πολλά ε, τα προβλήματα, οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα γνωρίζουν και ξέρουμε ότι είναι δυστυχώς... Ε, με την ε, νέα παγκόσμια τάξη πολλά τα προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. σε μια περίοδο αλλαγής, σε μια περίοδο ανάπλησης θα πρέπει ο καθένας, μια ομάδα, μια κοινωνία αλλά και όλα τα δικαιώματα των ε, πολιτών να ε, την χάνουν τις φροντίδες και τις μέρημνας των κυβερνήσεων και των κρατών. ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις, παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Υπάρχουν, πιστεύω, πέντε βασικά κεφάλαια ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η κοινωνία των πολιτών, η υπευθυνότητα και η δικαιοσύνη. Για να περάσουμε λοιπόν μέσα από μια διαδικασία μεταβατική θα πρέπει να ε, περάσουν ορισμένες χώρες από την ε, μετάβαση, από την ανάπλαση, από την αλλαγή μια αλλαγή, μια ανάπλαση την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει εξασφαλιστεί στην Τουρκία κατά τρόπο αρκετά επικοδομητικό, ουσιαστικό ή ταχύ. Πρόκειται για μια αδεξιότητα θα έλεγα που στην ε, Τουρκία σημαίνει ότι δεν υποστηρίζονται οι ε, δυναμικές εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή. Και έτσι Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει το δυναμικό, υπάρχει η βούληση για αλλαγή, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Ένα κύριο χαρακτηριστικό για την μετάβαση, για την ανάπλαση μιας κοινωνίας είναι η δικαιοσύνη. Είναι το να αντιμετωπίσει κατάματα το παρελθόν της, την ιστορία της. Σημαίνει μεγάλο θάρρος βεβαίως, μεγάλη παρησία εκ μέρους μιας κοινωνίας αυτό και σε μια χώρα όπως η Τουρκία που έχει πολλά, πολλές εθνότητες, πολλές διαφορετικές θρησκείες, ε, δόγματα, ε, είναι, απαρα... Ε, είναι ανάγκη να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να αποκαταστήσουμε την πληγωμένη δικαιοσύνη. Ωστόσο δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η ε, εργασία της μνήμης. Εμείς από την άλλη οι Κούρδοι που είναι ένας από τους λίγους λαούς που έχουν μείνει χωρίς κράτος δεν θέλουν να ξεχάσουν, δεν θέλουν να λησμονήσουν, θέλουν να μην πάνε οι θυσίες τους χαμένες. Έχουμε πολλές θυσίες, σφαγές, ε, εγκλήματα που έχουν για χρόνια ολόκληρα και δεκαετίες καταπληγή, Έχουμε την σφαγή του Ντέρσιν το 1938, τη ιστορικό πραξικόπημα το 1980, τα, την πραγματικότητα που ζουν οι κρατούμενοι στις φυλακές του Διάρμπακρ, του Μαμάκ, του Μετρίς. Έχουμε τη σφαγή του Χελέπτσε, του Ιράκ δηλαδή από τον ε, Σαντάμ Χουσέιν, τους ε, ομαδικούς τάφους, τους ε, φόνους που δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη, έχουμε τους αγνοούμενους, έχουμε πολλά εγκλήματα που δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε καταδίκες Όλα αυτά είναι πληγές που δεν έχουν γιατρευτεί. Και μάλιστα τα τελευταία επεισόδια στην περιοχή Τσουκούρτζα δείχνουν ότι το κράτος αποφασίζει να συνεχίσει την εμπόλεμη σχέση, την αντιμετώπιση των προβλημάτων σαν να ήταν μια εμπόλεμη κατάσταση. σε μια περίοδο μετάβασης χρειάζεται ένα ουσιαστικό μηχανισμός που θα διευκολύνει την απόδοση της δικαιοσύνης, την αναγνώριση της αλήθειας. Χρειάζεται λοιπόν θάρρος, χρειάζεται διορατικότητα, χρειάζεται βούληση, χρειάζεται σταθερότητα, ειλικρίνεια Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συναντήσεις μεταξύ των, της κυβερνήσεως του κράτους, δηλαδή του τουρκικού και του ΠΚΚ ε, και του Οτσαλάν, έχουν γίνει δεχτές από τον τουρκικό λαό με ε, πάντως όχι αντίδραση, όχι αρνητική αντίδραση. Πλην όμως ε, η κυβέρνηση του ΑΚΠ δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της έδινε η μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές και δυστυχώς αντί για τα θεμητά δικαιώματα των ε, Κούρδων, αντί για τα δίκαια αιτήματά τους, αντιμετωπίζουμε δεκάδες κρατήσεις, συλλήψεις, προσαγωγές και παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αντιμετωπίζουμε την κρατική τρομοκρατία. Και δυστυχώς ε, το να προτιμήσει κανείς να μείνει σιωπηλό σε μια τέτοια περίπτωση σημαίνει ταυτόχρονα και να πιστεύει ότι μπορεί κανείς να προτιμά μια να αποδέχεται μάλλον μια αθέμητη, μια άδικη, αρνητική πολιτική προπαγάνδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση με μια λεγόμενη τάμπουλα ράζα, με ένα από μηδενική ε, βάσεως νέο σύνταγμα. Ε, είναι κάτι το οποίο προχωρεί, πιστεύω, με πολλές προσδοκίες από πλευρά του λαού και με πολλή υποστήριξη. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάτι θετικό, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και την αντιμετώπιση του παρελθόντος. Πρέπει να μιλήσουμε για την αλήθεια, πρέπει να γίνουν οι δίκες, πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές αληθείας, πρέπει να υπάρξουν μουσεία, που είναι μερικά από τα παραδείγματα μόνο για την αναγνώριση του παρελθόντος. Υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη να προχωρήσουμε χωρίς περιορισμούς, όπως έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, στην αντιμετώπιση του παρελθόντος. Πρέπει πλέον να ανοίξουμε τα μάτια και να αναγνωρίσουμε την ιστορία μας. Αυτό σημαίνει για τους Κούρδους ιδιαίτερα αναζήτηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε φορά που κάποιος διεκδικεί το δικαίωμά του σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο Κούρδος δεν, είναι, δεν θα αναγνωρίζεται πλέον, δεν θα περιγράφεται πλέον ως ληστής, αλήτης, πλιατσικολόγος, ε, αποσχιστής ε, ή σήμερα τρομοκράτης σημαίνει ότι θα μπορέσει να βρει μια θέση στον κόσμο μέσα σε συνθήκες δικαιοσύνης, μια θέση μέσα στην επίσημη πολιτική και μια καθαρή τοποθέτηση η οποία θα μας επιτρέψει να ζήσουμε συνθήκες ειρήνης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Είμαι βέβαιος ότι θα ήταν εξίσου ευπρόσδεκτο το μήνυμα της κυρίας ε, Ζάνα και στα κουρδικά αν μας το διαβάζατε. Ο κύριος Κέλαμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι εκπροσωπώ την Εστονία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτος το οποίο δεν θα έπρεπε, εάν η ιστορία είχε πάρει το δρόμο της, να βρίσκεται σήμερα εδώ. Και γι' αυτό καταλαβαίνω πολύ καλά τα όσα είπατε. Εγώ είσαι επί 50 χρόνια της ζωής μου υπό δικτατορικό καθεστώς, στρατιωτική δικτατορία. Δεν ξέραμε τι σημαίνει ελευθερία, δεν ξέραμε τι σημαίνει να ορίζει κανείς το μέλλον του, τη μοίρα του. Ωστόσο, όπως είπατε κι εσείς και όπω είναι το θέμα του πάνελ μας, το αντικείμενο μας είναι μετάβαση στη δημοκρατία και νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς από την εμπειρία μας ε, μια ουσιαστική συμβολή για την πρόοδο προς τη δημοκρατία, την ελευθερία μάλλον και μια ουσιαστική δημοκρατία, μια όριμη δημοκρατία. Πάνω από όλα λοιπόν θα θέλω να πω ότι σημαντικό είναι να μην προσφέρετε στήριξη σε δικτατορικά καθεστώτα, να μην αποδέχεται κανείς τα επίσημα ψεύδη όπως έλεγε και νωρίτερα κάποιος, ας μην ζούμε μέσα στο ψέμα. Ας κρατήσουμε αποστάσεις από την επίσημη προπαγάνδα, από τα ψέματα. Και πρέπει να βοηθήσουμε στην οργάνωση της μετάβασης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί είναι πάντα δυνατόν αυτό. Υπάρχουν δυνατότητες να βοηθήσουμε τις παράνομες ομάδες, ε, τις εκτός νόμου ομάδες να ετοιμάζουν κείμενα, να οργανώνονται. Εγώ το 72 απέστειλα την πρώτη μου επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη και δεν περίμενα από τον Γενικό Γραμματέα κύριο Βάλτχάιμ να, να μου δώσει απάντηση. γιατί κυκλοφορούσε και η ιδέα ότι το 99,9% των Εστονών υποστήριζαν το ε, δικτατορικό καθεστώς του κομμουνιστικού μπλοκ. Ε, και έτσι μπορέσαμε να εκφράσουμε τη θέση ότι δεν ισχύει αυτό. Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας το 1978 ήμασταν προετοιμασμένοι, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και αυτό ήταν μεγάλο πλεονέκτημα και αρχίσαμε αμέσω να οργανώνουμε πρωτοβουλίες πολιτών. Με δημόσιες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, με συναθρήσεις δηλαδή, με την διαμόρφωση για πρώτη φορά πολιτικού κόμματος ε, στην Σοβιετική Ένωση, του εσθονικού Κόμματος της Ανεξαρτησίας, πολύ του τίτλου, και επίσης πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και ρόλο διαδραματίσαν οι πρωτοβουλίες των πολιτών, γιατί αποδεδειγμένα υπήρχε μια ευρύτατη πλειοψηφία των πολιτών πίσω από την ιδέα, πίσω από την διεκδίκηση για μια πραγματική και ουσιαστική ανεξαρτησία, όχι, πίσω από μια, όχι μια λυψή ε, ανεξαρτησία, αλλά μια ουσιαστική ανεξαρτησία ήταν αυτό που ζητούσαμε. Επίσης η λειτουργία των κομμάτων είχε πολύ μεγάλη σημασία. Οργανώσαμε μέσα σε ένα χρόνο πολλά πολιτικά κόμματα ταυτόχρονα μπορέσαμε να επηρεάσουμε και τις εργασίες του ε, αποδυναμούμενου πλέον Κομμουνιστικού Κόμματος και έτσι το 1989 όταν η επίσημη δικτατορία, το επίσημο δικτατορικό καθεστώς απεγνωσμένα προσπάθησε να αντιδράσει στις ε, πρωτοβουλίες μας ε, πλέον δεν ήταν αρκετά αποφασιστική, ήταν διστακτική το 1981 διορθώνω και έτσι δεν μπορούσε να αναλάβει πολύ αποφασιστικά δράση και με τον ε, πόλεμο στον Περσικό ο Γκόρμπατσοφ ε, προσπάθησε εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να καταστήλει τις ε, αντιδράσεις των πολιτών. Φτάσαμε στο 1991 όπου δεν γνωρίζαμε με τον πόλεμο τι μπορεί να προκύψει. Είμαστε όμως έτοιμοι να δεχθούμε κάθε ενδεχόμενο. Είναι εύκολο τώρα να πούμε ότι μπορέσαμε το 1991 να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των ε, βαλτικών κρατών, όμως δεν ήταν δεδομένο, δεδομένη αυτή η έκφαση πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι διατεθειμένος να αναλάβει κάθε προοπτική ως δεδομένη και κάτι μπορεί να προσφέρουν τα βαλτικά κράτη ως ε, ε διδασκαλία πιστεύω ότι δεν υπήρξε μίσος, δεν υπήρξε μυσαλλοδοξία, διάθεση για εκδίκηση και δεν έχασε τη ζωή του στα τέσσερα χρόνια της μετάβασης από το 87 μέχρι το 91 ούτε ένας ε, πολίτης. Μπορούμε λοιπόν ε, να σεμνινόμαστε ότι αυτή τη διαδικασία την ολοκληρώσαμε με αξιοπρέπεια κατά τρόπο ειρηνικό και δημοκρατικό. Και έτσι και έχουμε σήμερα καταφέρει και να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε μια πολύ υγιή, πρέπει να πω, δημοκρατία. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να έχουμε την υποστήριξη της εθνούς κοινότητας. Στην περίπτωση της Λιβύης, της Τινησίας, μπορούμε να διαπιστώσουμε και να καταγγείλουμε δυστυχώ τις συμφωνίες ντροπή με τους προηγούμενους, με τους πρώην δικτάτορες, με τους ε, Ανατραπέντε δικτάτορε και νομίζω ότι από αυτό πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα στην Ευρώπη. Θα πρέπει ή μη τι άλλο να σταθμίζονται τα οικονομικά συμφέροντα με αυτά που υπαγορεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Και κλείνοντα θα ήθελα να πω, εν προκειμένου, ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας ε, η ΓΟΜΕ έχει κάνει μια προσπάθεια για την ε, ε, διαμόρφωση του βραβείου Ζαχάροφ, διότι βλέπουμε ότι επικεντρωνόμαστε στη δραστηριότητα αυτή του βραβείου Ζαχάροφ περισσότερο τον Δεκέμβριο, με την απονομή δηλαδή. Όμως αυτό δεν ε, αντικατοπτρίζεται επαρκώς ε, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσο δεν έχει επαρκή απήχηση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσκαλεί κάθε και τους βραβευθέντες αλλά και τους υποψηφίους γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολη επιλογή κάθε χρόνο από τους πολυάριθμους ε, υποψηφίους που όλοι είναι εισάξιοι και αξίζουν να τιμηθούμε το βραβείο Ζαχάροφ να επιλέξουμε έναν. Πρέπει λοιπόν ε, να προσκαλούνται όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν στην Επιτροπή των ε, Εξωτερικών, στην Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε κάθε άλλη αντίστοιχη ή σχετική επιτροπή, ώστε να γίνεται αυτή η συζήτηση κάθε χρόνο. Για να μαθαίνουμε και εμείς ε, τι ε, μεσολάβησε τι συνέβη στη χρονιά που πέρασε ε, στη ζωή αυτών των ανθρώπων των τιμηθέντων με τον βραβείο Ζαχάροφ και σε τι έχουμε μπορέσει να βοηθήσουμε την κατάσταση. Και θα πρέπει να πω ότι η ιδέα μου περισσότερο είναι να, κάνουμε, να γίνουμε η πολιτική ανάδοχη αυτών των βραβευθέντων με το, ταμείο, με το βραβείο Ζαχάροφ. Δηλαδή να μην είναι άνθρωποι που απλώ τα καλούμε για να πονίμουμε ένα βραβείο μία μέρα, αλλά να είναι άνθρωποι που θα βρίσκουν ανοιχτή πάντα την ε, πόρτα μας, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και να έχουν μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια κάρτα πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορούν να, έρθουν, να έρχονται στα γραφεία μας. Η ΔΕ Υπηρεσία εξωτερική δράση και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπουδήποτε βρίσκονται και τώρα στα κράτη αυτών των τιμηθέντων με το βραβείο Ζαχάροφ θα πρέπει να διατηρούν ε, την επαφή μαζί του διαρκώ ώστε να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για τις συνθήκες διαβίωσης τους. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες αυτές και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τους βραβευμένους με το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι πολύ καλή ιδέα. Και με χαρά βλέπω εδώ και τον ε, Αλεξάνδερ και τη Λουτμίλα στην πρώτη σειρά. Κάποιος εκεί πίσω έχει ζητήσει το λόγο. 6 παρά 20 θα τελειώσουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μίριαμ Μπλακ. Είμαι ε, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΦΛΑ, που είναι η νομική αρρωγή για την Αφρική. Αλλά στην καθημερινή μου ζωή είμαι η πρέσβερα της Ουγκάντα. Θα ήθελα να εκφράσω θαυμασμό για όλους αυτούς τους θαραλέους βραβευμένους που έπαιξαν αυτό τον ρόλο στη χώρα τους προωθώντας ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ είμαστε σε ένα παγκόσμιο βήμα και θα ήθελα να συνταχθώ και εγώ με τα όσα είπε ο Σαλίος Μάν και η γραμματέας του Διεθνούς Δικαστηρίου για να δούμε ε, τι γίνεται με αυτούς τους πρώην δικτάτορες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. A country Ξέρετε τι έγινε ε, ε, με τον α, δικά μου δικτάτορα, ο οποίος ποτέ δεν πέρασε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είμαστε σε ειρήνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ουγγάντα γιατί ο Κόνη και οι στρατιώτες ε, έχουν απλώς καταφύγει στην χώρα της Κεντρικής Αφρικής όπως επίσης και στο Σουδάν και κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Δεν σκοτώνουν πια τους δικούς μας αλλά σκοτώνουν άλλους Αφρικανούς και απάγουν ε, κορίτσια για να τα υποδουλώσουν ε, σεξουαλικά. Θα πρέπει λοιπόν να υψώσουμε το ανάστημά μας και να εκφράσουμε με τη φωνή μας τα εκατομμύρια θύματα και να ζητήσουμε η διεθνής ε, κοινότητα να συνεργαστεί και να συλλάβει και να παραδώσει αυτούς τους εγκληματίες στο Διεθνέ Ποινικό ε, Δικαστήριο. Ξέρω πως έχει απευθύνει τέτοιες εκκλήσεις ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ρωτώ το πάνελ. Ξέρετε πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει αστυνομία δική του. Ίσως όμως κάποιοι εδώ στο πάνελ έχετε κάποιες ιδέες ή συστάσεις για το πώς μπορούμε αυτούς τους ε, εγκληματίες που έχουν διαπράξει τέτοια ή ε, ε, δεχθεί εγκλήματα στη δικαιοσύνη. Σε ένα λεπτό θα δώσω το λόγο στην Μπάρμπαρα να δώσει κάποια συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει στήσει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ. Στα γρήγορα για το τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μεταβατικές ε, περιόδους. Δεν θα πρέπει να, να παραβλέπετε τη σημασία που έχουν οι δικές σας επισκέψεις στις χώρες. Πολλά γίνονται στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλε, αλλά το πιο αποτελεσματικό είναι μία αντιπροσωπεία που πηγαίνει στη χώρα και δίνει συνεντεύξει τύπου στη χώρα. Μα το λένε πολύ συχνά. Ο αντίκτυπο είναι τεράστιο και όσο πιο συχνά ταξιδεύετε στι χώρε αυτέ, όσο πιο συχνά συναντάτε αυτού του υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο πιο πολύ βοηθάτε τη μεταβατική περίοδο. Και για του βραβευμένου, Είδα στην Πρίστινα τον ε, βραβευμένο μας ε, ε, από το Κωσυφοπαίδιο στην Πρίστινα. Αλλά δεν τον είδα ποτέ στο Κωσυφοπαίδιο. Είδατε λοιπόν τι μπορεί να κάνει το δικό σας βραβείο. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφράσετε σε όλες τις γλώσσες, ξεκινώντας με τα αραβικά, τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν είναι γνωστές. Γιατί λένε δεν κάνει τίποτα το Κοινοβούλιο, που είναι συνήθως εσφαλμένο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αναγνωστεί από όλους αυτούς τους ανθρώπους το έργο σας. Είναι λοιπόν κάτι εύκολο και πιστεύω πως α, αυτή η μετάφραση θα βοηθήσει των δικών σας θέσεων. Και για το πόσο ορατή είναι βραβευμένη με ε, βραβείο Ζαχάροφ, πιστεύω πως εκεί που βρίσκεται αυτός που έχει βραβευτεί, πιστεύω πως μια αντιπροσωπεία του βραβείου ε, Ζαχάροφ που θα επισκεφθεί την Λευκορωσία, την Κούβα ε, και που θα συνοδεύεται από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από ευρωβουλευτές, θα έχει τεράστια απήχηση. Uh, Εγώ πήγα στην Κούβα πρόσφατα και με τις μητέρες ε, με τα λευκά και με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους και πιστεύω ότι πραγματικά έχετε δίκιο. Αλλά γιατί θα δώσω στην Μπάρμπαρα Λόκουμπιλερ το λόγο που είναι πρόεδρος της υπό Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να, κάνει, ε, να μας δώσει τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο να συνθέσω αυτή την τόσο πλούσια συζήτηση. Βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δική μας πλευρά ε, θα ξανασυζητήσουμε κάποιες από τις ε, ιδέες, κυρίως ας πούμε αυτή τη δημιουργία δικτύου βραβευμένων με το βραβείο Ζαχάροφ. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μπεντσεντρίνη, η οποία είπε ότι χρειάζεται χρόνο και υπομονή η μετάβαση στη δημοκρατία. Ε, είναι ε, σωστό αυτό, άλλωστε είπε και ο κύριος ε, Βέστεντορπ, ότι δηλαδή δεν υπάρχει εγχειρίδιο που να μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο παντού και για όλους. Θα πρέπει να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η κάθε κοινωνία που βρίσκεται σε μετάβαση προς την δημοκρατία και βεβαίως οι ίδιες ε, οι κοινωνίες θα πρέπει να πάρουν ε, τις αποφάσεις τους. Ε, η κυρία Μπενσεντρίν μας θύμισε ότι η ίδια η κοινωνία στην Τινησία θα πρέπει να ασχοληθεί με την μετάβαση και να πάρει τις αποφάσεις. Σαφώς είπε ότι επιθυμεί για την Τινησία εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, έχει διαφανείς διαδικασίες απέναντι ε, στην ε, Τινησία. Ομοίως άκουσα και ότι χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να εισπράξουμε, να χωνέψουμε και να να αξιοποιήσουμε τα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτή τη μετάβαση. Βέβαια υπάρχουν πολλοί που υπεστήριξαν την οικουμενικότητα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της διεθνούς προστασίας που θα πρέπει να χαρακτηρίσει αυτήν την ε, ε, διαδικασία. Αυτό το ανέφερε Φερρυπίνη λέει Λαζάλα για την ανάγκη να συμπεριληφθεί η διαδικασία και η δικαιοσύνη μέσα στο νέο σύνταγμα. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρξει ατιμορρησία για εκείνους οι οποίοι μέσα σε μία κοινωνία ε, δικαιοσύνης και κράτους δικαίου δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αυτά τα βασικά δικαιώματα. Εσείς μιλήσετε πολύ ωραία κυρία μου λέγοντας νωρίτερα ότι πρέπει να απαλλακούμε από το φαρμάκι της δικτατορίας, από το δηλητήριο της δικτατορίας. Και επίσης και από την ιστορία της Τουρκίας με τα όσα ακούσαμε από την εκ μέρους μάλλον της Λέιλα Ζάνα βλέπουμε ότι χρειάζεται και να κάνουμε τη δουλειά της Αναγνώριση της ιστορίας και του παρελθόντος, της αντιπαράθεσης δηλαδή ε, με την ιστορία και το παρελθόν, πράγμα το οποίο μπορεί να κάνουν το Εθνικό Δικαστήριο, αλλά, ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και σε εθνικό επίπεδο, σε εσωτερικό επίπεδο. Δεν πρέπει δηλαδή ε, αυτά τα πράγματα να λησμονηθούν ταυτόχρονα, όμως δεν μπορεί κανείς αυτή την διαδικασία της αποκατάστασης να την αναπτύξει εμπνεόμενος από ε, πνεύμα μυσαλλοδοξίας, από πνεύμα εκδίκησης Ωστόσο πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιος ο οποίος είναι, ανήκει σε μια μειονότητα που έχει υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων του και καταπίεση πρέπει, έχει και το δικαίωμα της αποκατάστασης. Γι' αυτό σε κράτη όπως τα αφρικανικά πρέπει, ε, όπως είπατε και εσείς, να μην... φερόμαστε ε, αυτάρεσκα ή να επαναπαυόμαστε έναντι των δικτατόρων ε, των κρατών αυτών. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε δηλαδή τα καθεστώτα αυτά και προληπτικά να παρεμποδίζουμε την δραστηριότητά τους. Θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θες διατυπώσει ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση των διεθνών εγκλημάτων. Ε, μιλάμε δηλαδή για το διεθνές δικαστήριο και ξέρετε ότι έχει μεταφραστεί αυτό και στα αραβικά. Με πολλή λεπτομέρεια μπορείτε να διαβάσετε δηλαδή εκεί τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω και θα πρέπει οι δικτάτορες να προσάγονται στη δικαιοσύνη, αλλά ενώπιον εκείνων των οργάνων, εκείνων των δικαιοδοτικών οργάνων που έχουν σαν στόχο ακριβώς να εκδικάσουν τέτοιου είδους εγκλήματα και γι' αυτό καλούμε και τις μεγάλες χώρες και δυνάμεις του κόσμου να μην καταπολεμούν τα διεθνή δικαστήρια, να τα στηρίξουν. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει με τη Ρωσία, την Κίνα, αλλά σε έναν βαθμό και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η διαδικασία της μετάβασης, της μετάλλαξης σημαίνει ταυτόχρονα και επεξεργασία των, των ε, παραβιάσεων των ανθρωπινών δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί, να θυμόμαστε, να αναγνωρίσουμε και να προχωρήσουμε παραπέρα, να προχωρήσουμε προς τη δημοκρατία. Αυτό το ακούσαμε και από την Τινησία και από την Τουρκία. Ο κύριος Ζιάντε από την Συρία μας μίλησε πολύ ξεκάθαρα και μας περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα του λέγοντας ότι πολλοί είναι αυτοί που δεν φοβούνται πλέον ε, να ε, ξεσηκωθούν απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο έχει διαπράξει φόνους, το οποίο έχει βασανίσει, φυλακίσει τόσους πολλούς. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουν ξεπεράσει το φόβο πια οι άνθρωποι και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ρωτάμε πάντα τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να στηρίξουμε εκείνους οι οποίοι θέλουν να προαγάγουν αυτή την ε, μετάλλαξη. Το Κοινοβούλιο αυτό που μπορεί σίγουρα να κάνει να συζητά αυτά τα ζητήματα και όντως το πράττουμε, όντως τα συζητούμε για δε το αίτημα για την ε, επιβολή μιας ζώνης απαγόρευσης υπερπτήσεων ή για, την, για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων ή την στήριξη για μια ιδέα ουδέτερη ζώνη στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία πιστεύω ότι είναι κάτι στο οποίο βρίσκεται σε επίπεδο κοινοβουλίου Ευήκο ΑΟΤΑ. Ε, πρέπει πλέον να κάνουμε την προσπάθεια για να δεχθεί τις προτάσεις αυτές και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για την Κίνα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ε, πολύ στενά συνδεδεμένη οι συνθήκες οι οικονομικές με την ε, αποσιώπηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το είπε και ο κύριος Σκέλαν, το βλέπουμε και στα κράτη της ε, Βόρειας Αφρικής όπου γίνονταν ανεκτά τα εγκλήματα εις βάρος των πολιτών, τα βασανιστήρια, διότι θεωρούσαμε ότι είναι προς το συμφέρον μας να κρατήσουμε τα καθεστώτα αυτά ισχυρά, να είναι σφαλισμένα τα σύνορά τους, να μην μπορούν να περάσουν μετανάστες ή λαθρομετανάστες ή γιατί βρίσκονταν ε, σαν αλλακτική μόνοι ως υποψήφοι στην εξουσία Ισλαμιστές οι οποίοι δεν μας ήταν αρεστοί. Νομίζω ότι αυτά όλα καταγγέλλονται και στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορούμε να πούμε ότι πέραν αυτών των εγγράφων πρέπει να περάσουμε στην υλοποίηση. Τρίτο σημείο, η υποστήριξη και η ανάπτυξη κοινωνίας των πολιτών ενημερωμένης και δραστήριας. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια χώρα μεμονωμένη, όπως είπε και ο κύριος Σκέλα, να συνέβη στην ε, Εστονία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και μέσα σε μια διαδικασία μεταλλαγής πολύ ε, προηγμένη που σημαίνει, Φερρυπίνη για την Τινησία, ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της μετάλλαξης, της μετάβασης, είναι υπό επιτήρηση ή πρέπει να είναι ίσως υποτήρηση και μια νέα ενδεχόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ένα θέμα για την κυρία Τασλίμα Αναστρίν, που το υπογράμμισε ιδιαίτερος. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ε, σχετικοποίηση όσον αφορά το ε, θέματα νοοτροπιών, Φερρυπίν, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε πολύ συχνά το λάθος να μιλάμε για τις δυτικές αξίες. Λυσμονούμε ότι είναι οικουμενικές οι αξίες. Ακόμη και ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους είναι επίτευγμα που κερδίθηκε με πολλούς αγώνες στην Ευρώπη, με πολλή προσπάθεια, με πολύ ε, διαφωτιστικό έργο και σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι μία από τις θρησκείες ε, θρησκεία της πλειοψηφίας και ποτέ δεν είναι μία από τις θρησκείες θρησκεία της μειονότητας που ενδεχομένως θα υποστεί διώξεις. Αυτό ισχύει παντού. Και κλείνω με τα όσα είπε η κυρία Μπενζιτρίνε, η οποία ξεκάθαρα είπε πως ε, δεν είναι αντιφατικό να ζει κανεί σε μια μουσουλμανική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα ζει με βάση τις σύγχρονες αξίες, με τις οικουμενικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πιστεύω ότι όλοι μας εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές για σας και τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, Μπάρμπαρα. Ε, πραγματικά έκανες μια εξαιρετική σύνθεση όλων αυτών που ακούστηκαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ τους πανελίστε τους βραβευμένους, καθώς επίσης και τους βραβευμένους που δεν είναι παρόντες εδώ, για το θάρρος που έδειξαν, για τα όσα μας είπαν σήμερα εδώ. Και ευχαριστώ βεβαίως και όλους τους παριστάμενους ε, που ε, ήρθαν σήμερα εδώ, καθώς επίσης ε, και τις υπηρεσίες που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση. Η βραδινή μας συνάντηση ξεκινάει στις 19.30 στο Μποζάρ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.